Ich eröffne die Sitzung. Guten Tag, alle miteinander. Sie haben die Tages ναι, έχετε την ημερήσια διάταξη. Ε, έχει κανείς κάποια ένσταση, όχι. Ωραία, λοιπόν, έχετε τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης και θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι όπως συνήθως το τέλος της συνεδρίασης ε, αν θέλετε μπορείτε να υποβάλλετε κάποια ένσταση, κάποια παράπονα, αλλιώς ε, θεωρούνται ότι εγκρίνονται πρακτικά. Δεν έχουμε βουλγαρικά, τσεχικά, μαλτέζικα, σλοβένικα. Στη διερμηνία. Στην τελευταία τριμερή συνάντηση για το θέμα πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν αποκτηθεί μη κανονικά, μη, σύμφωνα με τον νόμο και συζητήσαμε ορισμένα πράγματα σε σχέση με το θέμα αυτό και η επόμενη ε, συνάντηση του Τριλόγου θα είναι στις, 8, στις 18 Φεβρουαρίου και φαντάζομαι ότι στο πλαίσιο της συνάντησης θα επιτευχθεί μια συμφωνία. Η κυρία Βεργιά ε, δήλωσε διατεθειμένη να περάσει μια συμφωνία και το Συμβούλιο επίσης δεν ήταν απρόθυμο τελικά να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας. Ω σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης έχουμε μια ανταλλαγή με τους εμπερογνώμονες για το θέμα των ευρωπαϊκών σχολείων. Και πάλι στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται το θέμα αυτό, για το οποίο έχουν εκπονηθεί ε, πολλά, πολλές εκθέσεις. Εγώ είχα συντάξει μια έκθεση δεκαετία του 90, ε, έχουμε μια έκθεση από την κυρία Χάνιμπαλ και από τον κύριο Ζαμαρί Καβαντάνη, τελευταία έκθεση. Επίσης καλέσαμε τον εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου που είναι το κεντρικό όργανο δείξει των σχολείων. Βεβαίω δεν μπορούσαμε να προσπαλέσουμε όλου του εκπροσώπου, γι' αυτό περιοριστήκαμε τέσσερι και συγκεντρωθήκαμε σε, σε ορισμένες χώρες που παίζουν σημαντικό ρόλο για το σύστημα αυτό. Βεβαίω δεν μπόρεσαν όλοι να παρευρεθούν, αλλά βρίσκονται εδώ, αλφαβητικά αναφέρω, η κυρία Σεσό Γκιμπέρ, που εκπροσωπεί το Ανώτατο Συμβούλιο τη Γαλλία, η κυρία Έλμπεκ που εκπροσωπεί την Γερμανία, ο κύριος Γκένιενς, την ε, φλαμανδική κοινότητα και η κυρία Ρομπά Χαμπιέ που εκπροσωπεί τη Γαλλία. Ε, το θέσαμε και πάλι ως μια ημερήσια διάταξη γιατί ε, τελικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι για το θέμα των ευρωπαϊκών σχολείων απευθύνονται σε εμά γιατί προφανώς υπάρχουν πολλές δυσλειτουργίες σε αυτά. Και επειδή στην ουσία δεν είμαστε εμεί αρμόδιοι ενώ όλοι θεωρούν ότι εμεί είμαστε αρμόδιοι και, και παρόλο που δεν γνωρίζω εγώ μέχρι τώρα ποιο είναι ακριβώς ο ρόλος μας, γιατί τελικά τα ψηφίσματά μας καταλήγουν στο καλάθι των αχρήστων. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλέσαμε ούτω ώστε να μας πείτε κάποια πράγματα ε, σε σχέση με το τι έγιναν οι συστάσεις μας και πολλές φορές ε, οι συνάδελφοι διατυπώνουν κάποιες συστάσεις που δυστυχώς ε, τελικά, όπως σας είπα, ε, πετιούνται. Το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων αυτών των σχολείων είναι αυτό το μυστηριώδες ανώτατο συμβούλιο και πραγματικά αναμένω με ανεπιμονησία να μου πούν οι ειδικοί τι ακριβώς κάνουν εκεί αλλά θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον κύριο Καβαντά, ο οποίος συνέδεξε τη τελευταία έκθεση και ο οποίος ε, αισθάνεται και αυτός εξίσου απογοητευμένος όπως και εγώ. Παρακαλώ κύριε Καβαντά. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα καλύψω τις ανησυχίες μου με τη χαρά που θα έχω να ακούσω πολλές διαφορετικές εθνικότητες να εκφραστούν ε, για αυτό το ζήτημα Παρά την τάση που προβάλλουμε να γίνουν τα ευρωπαϊκά σχολεία ένα υπόδειγμα εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη, ουσιαστικά το σύστημα εκπαίδευσης περιορίζεται σε μόλις 24.000 περίπου μαθητές. Χαμηλό αριθμό. Οι μαθητές των σχολείων αυτών είναι κυρίως παιδιά υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ε, στελεχών μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων 44% ε, βρίσκονται στα σχόλια αυτά και στο σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων οι μαθητές κατηγορίας 2 γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις συμφωνίες που έχουν συναυθεί μεταξύ των ε, σχολείων και ορισμένων οργανισμών και επιχειρήσεων. Εκπροσωπούν μόλις ε, το 5% των συνολικών μαθητών. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί και μάλιστα μετά την οικονομική κρίση. Για τα σχολεία των Βρυξέλλων, το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην υπογράψει πλέον συμβάσει κατηγορία Β. Όσον αφορά του μαθητέ κατηγορία 3, των οποίων οι γονεί πρέπει να καταβάλουν δίδακτρα, αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20% των μαθητών των ευρωπαϊκών σχολείων και αυτό το ποσοστό βρίσκεται σε μειωτική τάση ανησυχητική. Συνολικά λοιπόν έχουμε ένα σύστημα κλειστό. Από το από... Πολλοί θεωρούν τα σχολεία αυτά είναι ελιτίστικα παρότι αυτό δεν είναι ακριβές. Αλλά αντικατοπτρίζει μια άλλη πραγματικότητα, η, η, την ανάγκη του να πάνε σχολείο τα παιδιά ε, ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν σε χώρες ε, στις οποίες δεν ομιλείται η μητρική τους γλώσσα. Η έκθεση υιοθετήθηκε το 2011 και με ενδιαφέρον παρατηρώ ότι έχει αλλάξει τα τελευταία τρία χρόνια. Τι πράγματα έχουν βελτιωθεί και κατά πόσο οι διατυπώσεις αυτής της έκθεσης ε, αντικατοπτρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Τα κυριότερα προβλήματα που αναφέρονται και παραμένουν επίκαιρα είναι τέσσερες. τέσσερα. Πρώτα απ' όλα η χρηματοδότηση του συστήματος, δεύτερον η απόσπαση των καθηγητών, τρίτον ο υπερπληθισμός σε ορισμένα σχολεία, Βρυξέλλες, Λουξεμβουργό και Φραγκφούρτη, εκεί που υπάρχουν δηλαδή θεσμικά όργανα, Τέταρτον, η μεταρρύθμιση της δευτεροβαθμίας εκπαίδευσης και η πραγματική αξία του μπακαλωρέα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του συστήματος, υπάρχει έλλειψη αποσπασμένων καθηγητών. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί η κατανομή των χρηματικών δαπανών. Το σημερινό χρηματοδοτικό σύστημα φορτώνει υπερβολικά ορισμένα κράτη-μέλη πρέπει να ζητηθεί από το Ανατολικό Συμβούλιο να αναθεωρήσει το μοντέλο χρηματοδότηση των σχολείων και την πρόσληψη των καθηγητών. Η έκθεση αυτή παρατηρούσε επίση ε, ότι είναι ανησυχητική σε λήψει αποσπασμένου προσωπικού, διότι θα έπρεπε να αντισταθμιστούν με επιτόπου πρόσληψη διδασκόντων οι αμοιβέ των οποίων θα αναλαμβάνονταν από τα σχολεία. Σήμερα ο αριθμό των απασχολημένων καθηγητών είναι μόλι 1492 καθηγητές ε, ε, το 2061 που είναι υπεύθυνοι για μαθήματα οι επενδύσει των κρατών μελών μειώνονται υπέρ των ευρωπαϊκών σχολείων έτσι αποδεικνύεται κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με του αρμόδιου γνωρίζουμε την ιδιαίτερη κατάσταση των Βρετανών και των Ιρλανδών οι οποίοι για το αγγλικό τμήμα που είναι περίπου 5.000 μαθητές ε, πρέπει να παράσχουν καθηγητές ενώ ουσιαστικά οι δική τους υπηκότητας μαθητές είναι οι μισή μόλις. Θα έπρεπε λοιπόν να αποσπαστούν οι διπλάσιοι ε, διδάσκοντες από αυτούς που αντιστοιχούν στους πραγματικούς τους μαθητές πολλοί μαθητές ε, έχουν διαλέξει τα αγγλικά για τη γλώσσα σε αντίθεση με το 17% για τα γερμανικά και 23% για τα γαλλικά. Λυπούμαστε λοιπόν, που δεν συμμετέχουν οι Βρετανοί σε αυτή τη συζήτηση όπως και οι Ιρλανδοί, από όσο γνωρίζω εγώ. Δήλωσαν οι Βρετανοί ότι δεν πρόκειται να αποσπάσουν νέους καθηγητές, ούτε θα αντικαταστήσουν όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν ή να λήξει η σύμβασή τους. όλο το θέμα είναι πιο επίγον. Χρειάζεται διαρθρωτική προσέγγιση. Η συμβολή των κρατών μελών μπορεί να είναι απόσπαση καθηγητών που θα διδάσκουν στη μητρική τους γλώσσα, είτε χρηματοδότηση, χρηματοδοτική συμμετοχή, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη. Θα μπορούσαν επίσης να αποσπάσουν διδάσκοντες που θα διασφαλίζουν ε, διδασκαλία σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους γλώσσα παρότι αυτή η διατάξη έρχεται σε αντίθεση με τα όσα συνιστά η δική μου έκθεση όπου επέμνα ότι είναι σημαντικό η εκπαίδευση να παρέχεται από ανθρώπους ε, στη μητρική τους γλώσσα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων προέρχονται από δίγλωσσα οικογενειακά περιβάλλοντα στην πλειοψηφία τους και ότι αν οι καθηγητές τους μιλούν ε, τη γλώσσα τους ε, λιγότερο καλά από τη ίδια η οικογένειά τους, η αξιοπιστία των καθηγητών αυτών και γενικότερα του συστήματος υποβαθμίζεται. Διακυβεύεται. Να σας μιλήσω για τον προβολικό αριθμό μαθητών και το άνοιγμα του συστήματος. Η έκθεση υπενθύμησε ότι το άρθρο 1 της συνθήκης επέτρεπε σε άλλα παιδιά να φοιτούν στα ευρωπαϊκά σχολεία βάσει των όριων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και βάσει και των ε, κτίριων που υπάρχουν στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Ο αριθμός των κτηρίων αυτών ε, εμποδίζει το άνοιγμα των σχολείων σε περισσότερα παιδιά από τα παιδιά του προσωπικού των θεσμικών οργάνων. Τα σχολεία κυρίως στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο δεν είναι δυνατόν να ανοιχτούν με αυτόν τον τρόπο και έτσι οι μαθητές αυτοί βρίσκονται ουσιαστικά σε ένα περιορισμένο ε, σε περιορισμό ουσιαστικά δεν είναι δυνατόν για άλλα παιδιά να πάνε να φοιτήσουν σε τέτοια σχολεία εκτός των παιδιών των θεσμικών οργάνων. Αυτό ενισχύει τις προκαταλήψεις που ήδη είναι αρνητικές όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους υπαλλήλους. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για τη μετερρύθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βάσει της έκθεσης που εκπώνησα εγώ όπως και στην έκθεση του 2012 μπορούμε να διαβάσουμε το εξής το Σεπτέμβριο του 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση για το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων τα 50 σημεία του ψηφίσματος ε, εξετάζουν τις διάφορες πτυχές των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Το το Συμβούλιο σημείωσε τους προβληματισμούς όσον αφορά τα μέτρα που λήφθηκαν μετά από το ψήφισμα και έδωσε εντολή να υλοποιηθεί μια ομάδα εργασίας που θα ονομαστεί Οργανισμός Δευτεροβάθμιων Σπουδών για τον εξορθολογισμό των σπουδών και ειδικότερα για τα προαιρετικά μαθήματα. Η ομάδα εργασίας ε, κλήθηκε να συμπεριλάβει μια νέα δομή στις μελέτες του για τη δευτεροβαθμία εκπαίδευση με σκοπό μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα και για την οικονομική τύχη. Αυτά αναφέρονται εκεί. Οι γονείς ε, διαφώνησαν με την, προοπτική, με την προσπάθεια αναθεώρησης του συστήματος υπογράμμισαν ε, ότι οι μεταρρυθμίσεις ε, που προβλέπονταν υπήρχε κίνδυνος να καταλήξουν καταστάσεις όπου οι μαθητές θα μάθαιναν μαθηματικά σε μία γλώσσα, φυσική σε άλλη και χημεία σε μία τρίτη. Και ότι αυτές οι γλώσσες ε, μπορούσαν να αλλάζουν από το ένα έτος στο, στο επόμενο. Δηλαδή δεν θα υπήρχε συνέχεια και σαφής κατανόηση. Πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσουμε ότι η έκθεση επιμένει στη διεξαγωγή μελετών επιπτώσεων πριν από τη μεταρρύθμιση του συστήματος. Πρέπει να δούμε σε ποια κριτήρια βασίζεται η μεταρρύθμιση πριν αυτή ξεκινήσει. Πρέπει να δούμε πώς αξιολογείται η αξία του Ευρωπαϊκού Μπακαλωρέα, του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου σε σχέση με άλλα ε, πτυχία όπως το Διεθνές Μπακαλωρέα. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις αφού ακούσουμε όλους τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Κάποια πράγματα να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καβάντα για μια πραγματικά πλήρη διεξοδική έκθεση. Πολλά σημαντικά θέματα εμπεριέχει Πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι την απογοήτευση των περισσότερων. Τα πράγματα φαίνεται ότι επιδεινώθηκαν από τη δική μου έκθεση, δεν βελτιώθηκαν. Και πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε σε βάθος πού πηγαίνουμε με τα ευρωπαϊκά σχολεία, ποια κατεύθυνση ακολουθούμε, πώς θέλουμε να λειτουργούν. Και να εξετάσουμε τα τέσσερα σημεία, τα τέσσερα θέματα ως άξονες που ανέφερε ο κύριος Καβαντά και απόλυτα συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχουν μελέτες επιπτώσεων, αξιολογήσεις επιπτώσεων. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα είδους σχόλιο. Σε σχέση με την έκθεσή μου αυτό ήταν ένα θέμα. Τα, τα αγγλικά είναι πολύ περισσότερο η γλώσσα σήμερα στο σχολικό σύστημα σαν αποτέλεσμα της διεύρυνσης. Και πάντα είχαμε ένα πρόβλημα με αυτό, υπήρχε πρόβλημα με αυτό τοπικό πρόβλημα σε σχέση και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι συμβαίνει, εμεί χρησιμοποιούμε τοπικά δασκάλους στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με αυτούς που προσλαμβάνουν οι τοπικές αρχές ε, παιδείας και εκπαίδευσης. Ε, κάπως αλλάζουν τα πράγματα τώρα. <clears throat> Δεν απασχολούνται από την ε, κεντρική κυβέρνηση με συμβάσεις και συμβόλαια. Πράγμα το οποίο κάνει αυτή την πτυχή πιο δύσκολη. Ακόμα και αν θέλουν ε, να πάνε σε σχέση με αυτό το εγχείρημα για 5 ή 7 χρόνια, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα μετά ότι δεν θα βρουν θέση απασχόλησης όταν θα επιστρέψουν από εκεί που ξεκίνησαν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί, γιατί δηλαδή δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί που να υποβάλουν αιτήσει και να θέλουν να συμμετάσχουν. Δεν ξέρω ακριβώς τα στοιχεία σχετικά, όμως αυτό είναι πάντα ένα θέμα σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό φαίνεται ότι επειδή Ενώθηκε σημαντικά ακόμα και συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση σε μια άλλη γλώσσα. Για, αυτά, για τους λόγους που προανέφερε ο κ. Καβαντά. Και αυτό πιστεύω ότι ουσιαστικά πρέπει να το συζητήσουμε εκτενέστερα με τις αρμόδιες αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο και, ε, και την Ιρλανδία. Να δούμε τι γίνεται, πώς θα επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Καβαντά. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης στην μητρική γλώσσα ενός ατόμου. Όχι ε, δύσκολο, αλλά καταλαβαίνω σε σχέση με τους ε, διερμηνείς ε, και τη δουλειά που κάνουν. Όμως καμιά φορά όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα έλεγε ο, ο ντόπιο, ο γηγενή. Τώρα και σε σχέση με τα παιδιά όταν τα διδάσκουμε πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Η γλώσσα στην οποία διδάσκονται πρέπει να είναι πραγματικά να μπορούν να μαθαίνουν από κάποιον που έχει τη γλώσσα αυτή ως μητρική γλώσσα, από κάποιον που μιλάει τα αγγλικά ως μητρική γλώσσα. Μπορούμε να βρούμε τέτοιους ε, ανθρώπους, ε, αλλά είναι σημαντική η αρχή του να είναι μητρική η γλώσσα τους. Πρέπει να το δούμε αυτό, πώς θα αντιμετωπιστεί Κάποια από αυτά τα προβλήματα συνδέονται και με τους μισθούς και τη χρηματοδότηση και το πώς δηλαδή χρηματοδοτούνται αυτά τα εγχειρήματα και υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε σχέση με αυτά τα κονδύλια και επιπρόσθετα έχουμε και το θέμα των ε, ε, διευκολύνσεων εγκαταστάσεων και ε, σε σχέση με τη δική μου έκθεση είχαμε θέματα τα οποία αντιμετωπίζαμε που φαίνεται ότι επιδεινώθηκαν και σημαντικά κιόλας από τότε μέχρι σήμερα. Γινόταν ε, λόγος ε, για να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, οι κατάλληλες δυνατότητες. Δεν έχουν επιληθεί όλα αυτά. Και θα ήθελα επίσης στο τέλος να μιλήσω και για το curriculum, τα μαθήματα χρειάζονται αξιολογήσεις ε, για το τι γίνεται και τι διδάσκεται. Και πάλι είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει για την αξία δηλαδή του ευρωπαϊκού μπακαλωρεά, του ευρωπαϊκού απολυτηρίου και μήπως ε, θα έπρεπε να υπάρχει η δυνατότητα ενός εθνικού απολυτηρίου ίσως. Και τώρα όλα αυτά εμεί προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε να βελτιώσουμε τα ευρωπαϊκά σχολεία σε αυτά τα πλαίσια και για κάποιους λόγους δεν προχωράμε. Θα έλπιζα και ελπίζω ότι δεν θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα και γιατί διαφορετικά θα υποβαθμιστούν τα ευρωπαϊκά σχολεία σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε πως ε, λειτουργούσαν στο παρελθόν και αυτό θα είναι αρνητικό. Λυπούμε που ακούγομαι κάπως απογοητευμένοι, υπάρχει κάποια απεσιοδοξία στις παρατηρήσεις μου. Υπάρχουν όμως πολλά θέματα τα οποία επιδεινώνονται, επιδεινώθηκαν και πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν. Ευχαριστώ. Tja, jetzt haben wir Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Έχουμε του Ανώτατου Συμβουλίου εδώ. Δεν έχουμε κανένα από το Ηνωμένο Βασίλειο όμως. Τις επόμενε ημέρες κάτι θα μας αποστείλουν. Αλλά σήμερα έχουμε του συναδέλφους εδώ παρόντες και παρούσες που γνωρίζουν αυτά τα προβλήματα και έχουν εξοικειωθεί με την κατάσταση. Θα ήθελα να μάθουμε κάτι για τα κριτήρια της χρηματικής, χρηματοδοτικής συμμετοχή των χωρών, cost sharing και να ξέρουμε τι γίνεται σε σχέση με την συμφωνία ε, σε σχέση με τη συμφωνία Σίφστατ ε, τι κάνει το Βέλγιο για παράδειγμα είναι πράγματα τα οποία από την κυρία Ρομπερ Μπαρμπιέ θα μπορούσαμε να ακούσουμε αν είχατε τη δυνατότητα να απαντήσετε και να τοποθετηθείτε παρακαλώ κυρία Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση, παρακαλώ, γιατί δεν περίμενα να μου δώσετε το λόγο τόσο γρήγορα. Ναι, μεταξύ άλλων cost sharing, η συμμετοχή στη χρηματοδότηση από πλευρά των χωρών. Τι φαντάζεστε τι πρέπει να γίνει με την έδρα κράτους. Ε, πώ αντιμετωπίζετε το θέμα της έδρα από το Βέλγιο. Ένα πέμπτο ευρωπαϊκό σχολείο θα ε, εγερθεί, θα ιδρυθεί. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα. Ίσως μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για αυτά παρακαλώ. können Sie auch an Herrn Gentjes weitergeben, aber ich denke... Αλλά μπορείτε να δώσετε το λόγο στον κύριο Γκέντζιες, αλλά νομίζω μπορείτε να απαντήσετε εσείς, θα γινόταν αυτό. Je pense aussi, mais je pense que vous... Πιστεύω, αλλά νομίζω ότι έχετε κάνει πολλές ερωτήσεις ταυτόχρονα. Είναι λοιπόν δύσκολο να τις απαντήσει κανείς όλες μαζί. Δεν ζήτησε το Βέλγιο πέμπτο σχολείο, το Ανώτο Συμβούλιο ζητάει πέμπτο σχολείο στις Βρυξέλλες όσον αφορά τον καταμερισμό του κόστου, Αυτή η απόφαση πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο ανώτου του Συμβουλίου. Λοιπόν, ζητάτε τώρα να πάρει το Βέλγιο θέση, αλλά αυτό δεν γίνεται. Καλύτερα να δώσουμε το λόγο στο Γενικό γραμματεία του Ανώτου του Συμβουλίου, που βρίσκεται σε καλύτερη θέση να σας πει πώς απάντησε το Ανώτο Συμβούλιο με το δικό του τρόπο στην έκθεση Καβάντα. Νομίζω ότι ανήκατε στο Ανώτατο Συμβούλιο και το Ανώτατο Συμβούλιο ήθελε να ηγεθεί αυτό το σχολείο. Αυτό σα ρώτησα. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε εσεί, ο κύριο Γκέντσιε μπορεί να πει κάτι. Um, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά δεν είναι κάτι απλό. Όπως θα έχετε αντιληφθεί, τίποτα στο βελίο δεν είναι απλό αφού μας ε, συστήσατε ως εκπροσώπους του Ανώτου Συμβουλίου των ε, Γλωσσικών ε, Κοινοτήτων του Βελγίου. Ουσιαστικά όσον αφορά την οικοδόμηση των σχολείων, το Ομοσπονδιακό κράτος του Βελγίου είναι αρμόδιο γι' αυτό. Όπως νομίζω, από πολλούς συναδέλφους, ανησυχούν ιδιαίτερα και ασχολούνται επισταμένα με το φάκελο αυτό. Θα γνωρίζετε επίση ότι φέτο είναι χρονιά εκλογών. Μια τέτοια χρονιά δεν είναι ποτέ καλή για να λαμβάνονται αποφάσεις τόσο σημαντικές όσο αυτή. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Νομίζω ότι ήταν πολύ ευαίσθητο το σύστημα, αλλά δεν είναι. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατό, αλλά προ το παρόν δεν έχουμε να σα πούμε κάτι παραπάνω. Συγγνώμη που δεν μπορώ να σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε. Τώρα, όσον αφορά το cost sharing, ναι, πρέπει να σα πω το ίδιο όπω ο συναδελφό μου. για αυτό το θέμα αποφασίζει το Ανώτο Συμβούλιο. Ψηφίζουμε εμείς ε, ατομικά φυσικά, αλλά δεν μπορώ να σας πω μια ατομική άποψη. Ε, υποστηρίζουμε εντελεί αυτό που αποφασίζεται τελικά από το Ανώτο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί σας προσκαλέσαμε τότε αφού δεν μας λέτε κάτι. Το Ανώτατο Συμβούλιο αποτελείται από ατομικά μέλη. Ατομικά από κάποια μέλη. Συλλογικά ίσως αποφασίζουν αλλά από εσά ατομικά αναμένω να μας δώσετε τις δικές σας απόψεις. Ποιες είναι οι δικές σας απόψεις για το cost sharing. Δεν θέλω να μου δώσετε εσείς κομμένη και ραμμένη την ε, νομική πράξη, αλλά πώς φαντάζεστε εσείς προσωπικά ότι θα έπρεπε να διαμορφωθεί το cost sharing. Ποιον να ρωτήσω. Το Ανώτατο Συμβούλιο δεν είναι ένα άτομο, είναι αρκετά διαφορετικά άτομα. Και ρωτώ εσείς, ο άλλος, ο παρά ποια είναι η άποψή σας. Σκεφτείτε ίσως τι μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα. Κανείς από τους άλλους συναδέλφους να δώσει εδώ κάποια απάντηση. Ε, ευχαριστώ. Ε, και αυτή ήταν μια απάντηση. Ίσως η κυρία Σασό Γκιμπέρ θα μπορούσε να μας ε, δώσει την άποψή της. Γιατί τα γαλλικά εκπροσωπούν το μεγαλύτερο τμήμα. Έχετε 6.000 ενώ στα αγγλικά είναι 5.000. Ίσως θα μπορούσατε λοιπόν εσείς να μας πείτε τι γίνεται στη Γαλλία με την απόσπαση τον του δακτικού προσωπικού ή θα μπορούσατε να απαντήσετε την ερώτηση του κυρίου Καβαντάη σε μια παρατηρήση της κυρίας Χάνιμπαλ. Ε, δεν χρειάζεται να φέρετε σε μένα, άλλωστε υπόθηκαν τόσα πολλά που ε, κατ' θα μπορούσατε να δώσετε τη μία ή την άλλη απάντηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Χαιρόμαστε που ήρθατε, ίσως θα μπορούσατε να μας απαντήσετε και κάτι κυρία Σοζό. Mm, um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλη ευχαρίστηση θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Να σου πω πρώτα απ' όλα ότι η Γαλλία υποστηρίζει ιδιαίτερα τα ευρωπαϊκά σχολεία για την αξία του την αξία της πολυγλωσσίας, τι πολυπολιτισμικές αξίες αλλά και τι δημοκρατικές αξίες. Τα σχόλια αυτά έχουν περιοριστεί στις 28 το Ανωτού Συμβούλιο συνεδριάζει δύο-τρεις φορές το χρόνο με πολύ ωραίες ε, συναντήσεις και εκεί διαβουλευόμαστε με τρόπο δημοκρατικό και αρκετά αυστηρό. Υποστηρίζουμε στεναρά τις θέσεις μας που είναι θέσεις κρατικές, εθνικές, αλλά τα πράγματα δεν λαμβάνουν χώρα μόνο σε αυτές τις συνεδριάσεις. Συνεργαζόμαστε στενά με το Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Γίνονται ανταλλαγές για τις ομάδε εργασία, για τους διάφορου ελέγχους και οι ανταλλαγές αυτές γίνονται καθημερινά. Με τη μέρη να, να εξελιχθούν μαζί όλα αυτά τα σχολεία, να δημιουργηθεί αυτή η οδός που ακολουθούμε για να αποδείξουμε ότι αυτά τα σχολεία μετά τα 50 χρόνια ύπαρξή τους παραμένουν ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα που βρίσκεται πάντα μπροστά από όλα τα υπόλοιπα και που αντικατοπτρίζει τις παιδαγωγικούς μας σκοπούς. Η Γαλλία θέλει να υποστηρίξει, υποστηρίζει την εξέλιξη των σχολείων αυτών, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι ο Υπουργό Περού φέτος αποφάσισε το Σεπτεμβρίο να συμμετάσχει με περισσότερους διδάσκοντες και για την πρωτοβαθμία και δευτεροβαθμία εκπαίδευση ώστε να δείξει σε αυτές τις δύσκολες εποχές ε, τη βούληση για τέτοια επένδυση. Πέραν από τη δημιουργία θέσεων εργασίας αυτών, ε, μίλαμε και για Γάλλους επιθεωρητές, ε, επιθεωρητές παιδείας, και με, θα φροντίσουμε να βρούμε στη Γαλλία τους καλύτερους από τους καθηγητές και επιθεωρητές μας ώστε να τους αποσπάσουμε στα σχολεία αυτά και να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τα σχολεία αυτά. Υπάρχει λοιπόν για τα σχολεία αυτά μια πραγματική πολιτική στη Γαλλία με καθημερινή δέσμευση αλλά και με υψηλή ποιότητα διαχείριση του προσωπικού για το καλό των μαθητών. Αυτά είχα να σας πω όλα τα σημερινά μοντέλα που έχουν παρουσιαστεί τα διορθωτικά μοντέλα Απορρέωνα από τους προβληματισμούς των ομάδων εργασίας για το cost sharing ε, τα έχει ψηφίσει η Γαλλία, τα έχει υπερψηφίσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην παρουσιαφάση φάση θεωρώ ότι έχω απαντήσει σε ερωτήσεις σας. Ε, Φανώς η απόσπαση από τη Γαλλία είναι πιο εύκολη από την Αγγλία γιατί η Γαλλία είναι ένα συγκεντρωτικό κράτο και στο βαθμό αυτό είναι πιο εύκολο να αποσπαστεί το διδακτικό προσωπικό. Τα προβλήματα τα οποία περιέγραψε η κυρία Χάνιμπαλ υπάρχουν σε κάθε ομοσπονδιακό κράτο, όπω και στη Γερμανία επί παραδείγματα. Κυρία Έλμπεκ, θα ήθελα να σας δώσω σε εσά τώρα το λόγο για να μας πείτε πώς είναι η κατάσταση στη Γερμανία. Γιατί και εκεί υπάρχουν κενές θέσεις και αφορούν βεβαίως τους ε, γερμανόφωνους διδάσκοντες. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κάποια πράγματα για την κατάσταση της γερμανικής γλώσσας και, την, ε, και πώς γίνεται η διδασκαλία της στα ευρωπαϊκά σχολεία. Παρακαλώ κυρία Άλβερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Από όσο γνωρίζω, γερμανικές θέσεις, ε, δεν υπάρχει πρόβλημα να να βρεθεί προσωπικό. Δεν είναι κενές. Εγώ η ίδια δεν είμαι μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου. Ίσως μου έχουν διαφύγει κάποιες πληροφορίες, αλλά από όσο γνωρίζω δεν μένουν κενές ε, θέσεις γερμανικών στα ευρωπαϊκά σχολεία ε, και σε σχέση με αυτό που γίνεται στη Φραγκφούρτη όπου είναι πλεονάζον το προσωπικό, αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε και προηγουμένως το θέμα των κτηριακών υποδομών για τα σχολεία, όπου πράγματι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μόνο ε, λόγω της ε, μεταφοράς της ε, εποπτείας των τραπεζών στη Φραγκφούρτη Έχουμε προβλήματα με τα ευρωπαϊκά σχολεία όσον αφορά το δυναμικό τους ε, και προσπαθούμε να βρούμε μέσω και μακροπρόθεσμα κάποιες λύσεις, κάτι το οποίο είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Στη Φραγκφούρτη δεν έχουμε μόνο ένα σχολείο τύπου 1, δηλαδή το σχολείο στο Μπράουνχάιμ, αλλά έχουμε επίσης και ένα σχολείο στο Μπατ Φίλμπελ, ένα αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό σχολείο δηλαδή, το οποίο έχει τον αντίστοιχο δυναμικό και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε το ε, τι θα γίνει με τα παιδιά που θα μας έρθουν γιατί ε, θα είναι πλεονάζουν ο αριθμός των παιδιών και δεν μπορούμε να τα φιλοξενήσουμε στο σχολείο. Το σχολείο στο Μόναχο και αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό σχολείο λέει η κυρία Πάκα, εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα. Στο Μόναχο ε, Εκεί φροντίζει για τα κτίρια το, η κεντρική κυβέρνηση. Στη Φραγκφούρτη ήταν ε, το Ομόσπονδο Κρατήδιο. Ε, στο Μόναχο υπάρχουν κάποιες ε, καθυστερήσεις, ε, αλλά είναι άλλου είδους ε, τα προβλήματα και υπάρχει και μια ειδική ρυθμίση για τη χρηματοδότηση εκεί. Ευχαριστώ πολύ. θέλει κανείς από τους εκπροσώπους του Ανατάτου Συμβουλίου που είναι παρόντες να αναφερθεί σε κάποια από τα προβλήματα τα οποία έθεσε ο κύριος Καβαντά ή δεν θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο. Παρακαλώ. My name is Kari Kivinen, I'm the Secretary General. Το όνομά μου είναι I'm the Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων, εκπροσωπώ το Ανώτο Συμβούλιο εκτός των συνεδριάσεων του Ανώτου Συμβούλιο και έχω ετοιμάσει ένα μικρό PowerPoint για σας, εάν θέλετε να το δείτε. Μπορώ να το περάσω πολύ γρήγορα, δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσουμε στον κύριο Καβαντά στα όσα είπε και μετά να εστιάσουμε περισσότερο τι συζητήσεις μας στα προβληματικά σημεία όπως τα βλέπουν τα μέλη του Ανώτου Συμβουλίου. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξω θέση. Το Ανώτο Συμβούλιο λοιπόν έλαβε την έκθεση Καβαντά που συζητήθηκε στη συνάντηση στην Οξφόρδη το 2012. Σχολιάστηκε με σημεία δράσης. Πολλές δράσεις σχεδιάστηκαν βάσει της έκθεσης Καβαντά. Θα σας τα παρουσιάσω σημείο προς σημείο, τμήμα προς τμήμα, εν συντομία. Θα σας παρουσιάσω τα ίσω έχουν γίνει. Ο κύριος Καβαντά ανέφερε ότι πρέπει να ανοίξει το Ευρωπαϊκό Μπακαλωρέα και αυτό ακριβώς πράξαμε. Το Ευρωπαϊκ... Οι κανόνες του Ευρωπαϊκού Μπακαλωρέα μεταρρυθμίστηκαν ώστε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά σχολεία να μπορούν να προσφέρουν το Ευρωπαϊκό Μπακαλωρέα πέραν των 40 υπαρχόντων ευρωπαϊκών σχολείων. Υπάρχει λοιπόν σήμερα η δυνατότητα αυτή. Για παράδειγμα, πέρσι το καλοκαίρι είχαμε δύο διαπιστευμένα σχολεία που προσέφεραν το Μπακαλωρέα για πρώτη φορά στο Ελσίνκι και στο Μανόσκ και του χρόνου θα αποφυτίσουν οι πρώτοι αποφυτοί από το Ευρωπαϊκό Σχολείο του Στρασβούργου. Είναι λοιπόν μια διαδικασία σε εξέλιξη, συνέστησε ο κ. Καβαντά, τα ευρωπαϊκά σχολεία να μην είναι κλειστά, να τα ανοίξουμε περισσότερο, βάσει της σύσταση και της συνεργασίας με τη γαλλική αντιπροσωπεία και την ομάδα εργασίας ε, που είναι αρμόδια για το άνοιγμα του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων, ανοίξαμε πολλά νέα διαπιστευμένα ευρωπαϊκά σχολεία μετά από την εκθέση του κ. Καβαντά. Μπορείτε να δείτε εδώ τον κατάλογο. Και εγώ έρχομαι τώρα από τη συνάντηση των επιθεωρητών που συζητήσαμε το νέο σχολείο του Μπρίντιζη στην Ιταλία. Δέκα χώρες περιμένουν για να ανοίξουν ευρωπαϊκά σχολεία. Και διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή με αυτές. Το επόμενο θα είναι στο Ζάγκρεμπ. Και έχουμε και την χώρα, την Κροατία, που θέλει Ευρωπαϊκό Σχολείο στην επικράτειά τη. Εκδηλώνεται λοιπόν τεράστιο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά σχολεία και το δίκτυο των ευρωπαϊκών σχολείων διευρύνεται διαρκώ. Ο κ. Καόντα έκανε μια παρατήρηση ότι η αυτονομία των σχολείων πρέπει να γίνει ευρύτερη. Ε, Πολλέ αποφάσει έχει λάβει το Ανώτο Συμβούλιο όπου τα διοικητικά συμβούλια των σχολείων, όχι οι διευθυντέ, έχουν περισσότερε εξουσίε λήψη αποφάσεων. Στα διοικητικά συμβούλια συμμετέχουν οι γονεί, οι καθηγητέ, τα μέλη του προσωπικού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ανώτο Συμβούλιο, η Γενική Γραμματεία. Όλοι αυτοί αντιπροσωπεύονται στα αυτά τα διοικητικά συμβούλια των σχολείων. Τώρα, όσον αφορά τα ε, διδακτικά βιβλία. Μεταρρυθμίζονται μόνιμα. Μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα μα και να δείτε ότι όλα μα τα διδακτικά βιβλία για όλα τα θέματα από το νηπιαγωγείο μέχρι το τελευταίο έτος στον Μπακαλωρεά αναθεωρούνται κάθε δύο χρόνια. Ε, δύο ή τρία εκκρεμούν αυτή τη στιγμή και βρισκόνται υπό συζήτηση μέσα στις επόμενες εβδομάδες στην κοινή διδακτική επιτροπή. Αυτή την εβδομάδα για παράδειγμα μόλις ε, δεχτήκαμε, αναθεωρήσαμε, ε, λαμβάνουμε αποφάσεις για εννιά διδακτικά βιβλία όπως τα ICT, λατινικά, ελτρία, γεωγραφία, λετωνικά κτλ. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το πρόγραμμα σπουδών μας που θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα για πολλά άλλα εθνικά συστήματα. Πρόκειται πραγματικά για ένα δημιουργικό και ενδιαφέρον έργο το οποίο φαίνεται πρακτικά να εφαρμόζεται με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο κ. Καβαντά ονόμασε το νομικό μας καθεστώς ως αβέβαιο στην έκθεσή του και εμείς προσβληθήκαμε κάπως Παρ' όλα αυτά, το μελετήσαμε, το εξετάσαμε και διαπιστώσαμε ότι πράγματι πρέπει να βελτιώσουμε την νομική προστασία των καθηγητών, των γονέων, των μαθητών μας, των μελών του προσωπικού μας. Το Ανώτο Συμβούλιο λοιπόν να συζήτησε το νομικό καθεστώς σε δύο συνεδριάσεις και δεν υπάρχει τώρα μια ομάδα εργασίας νομικής προστασίας με μέλη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωπο των κρατών μελών. Όλοι αυτοί συζητούν το μελλοντικό νομικό καθεστώ των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή η συνθήκη, διότι είναι αρκετά περιοριστική όσον αφορά αυτή την επιλογή και αυτή την τύχη. Προτάθηκε να διεξαχθεί εξωτερική μελέτη όσον αφορά τα παιδαγωγικά αποτελέσματα που έχουν οι μαθητές μας. Έκτοτε εξετάζουμε τις δυνατότητες συμμετοχής σε ανεξάρτητες μελέτες, διεθνείς μελέτες και τις δυνατότητες συμμετοχής στο πιλωτικό έργο ε, πίσα του ΟΣΑ. Συμμετείχαμε εκεί λοιπόν. Τα αποτελέσματα με το σχολείο του Καλχάμ και τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. 15χρονοι μαθητές ε, είχαν επιδόσεις από τις καλύτερες στον κόσμο. Μπορείτε να κατεβάσετε από το διαδίκτυο τη μελέτη. Υπάρχει μια στοσελίδα όπου μπορείτε να την κατεβάσετε από τον ΩΣΑ. Πέραν αυτού συμμετείχαμε και σε άλλες ε, μελέτες ε, πίσω, για παράδειγμα στο Λουξεμβούργο και επικυρώθηκαν εκεί, βεβαιώθηκαν αυτά τα αποτελέσματα. Αναμένουμε τώρα τα αποτελέσματα ε, του δεκμών πίσω για το σχολείο του Λουξεμβούργου. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καβαντά όσον αφορά τη δύσκολη κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Έχουμε 450 υπεράριθμους μαθητές κάθε χρόνο. Που οφείλεται απλά στην ευρωπαϊκή διεύρυνση και στην ε, εξέλιξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και στις δυνατότητες του Βελγίου να χτίσει περισσότερα σχολεία. Είναι εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση την παρουσία να σας δώσω μια γενική εικόνα και μιλώ τώρα μόνο για τα σχολεία των Βρυξελών. Ανοίξαμε το νέο σχολείο στο Λάκεν πέρυσι, το 2012, το Σεπτέμβριο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.000 μαθητές και υπολογίζουμε ότι θα είναι πλήρες μέσα σε δύο χρόνια. Ζητήσαμε τη βελική κυβέρνηση να μας χτίσει ένα πέμπτο σχολείο και πρέπει να πω ότι ήταν πολύ θετικέ οι διαπραγματεύσεις με τη γαλλική και με τη φλαμανδική κοινότητα μαζί με ε, την αντιπροσωπή του Βελγίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνήσαμε για τους αριθμούς, για τις ανάγκες, για το χρονοδιάγραμμα και σύμφωνα με τη συμβαστική μας συμφωνία χρειαζόμαστε χίλιες σχολικές θέσεις μέχρι το 2015. Αυτό μπορεί να γίνει εάν ε, το Συμβούλιο Υπουργών ε, του Βελγίου συμφωνήσει να μας δώσει τα κτίρια στον Μπαρκεντάλ. Χρειαζόμαστε ένα πλέον σχολείο για 1.500 μαθητές το 2019 και αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με τις βελικές αρχές ε, τον τόπο και το χρονοδιάγραμμα του έργου αυτού. Αλλά χρειαζόμαστε κάποια πολιτική απόφαση, όπως υπόθηκε και από τους Βέλγους συναδέλφους μας. Και πάλι συμφωνώ απόλυτα με την έκθεση του κ. Καβαντά όσον αφορά τον προπολογισμό. Ήταν πολύ δύσκολα τα τελευταία δημοσιονομικά χρόνια. Γιατί? Διότι ο αριθμό μαθητών κατηγορία 1 που δεν ουσιαστικά καταβάλουν κανένα, καθόλου διδάκτρα αυξάνεται. Ο αριθμό των ε, μαθητών κατηγορία 2 και 3 μειώνεται. Διότι ο χώρο καταλαμβάνεται από μαθητέ κατηγορία 1 αλλά και επίσης λόγω της κρίσης στα κρατημέλη. Σε πολλές χώρες ο τομέας της παιδείας είδε περικοπές στους μισθούς και αυτό επηρεάζει άμεσα και εμάς. Έτσι λοιπόν έχουμε λιγότερα έσοδα από τα 28 κρατημέλη από ό,τι είχαμε προβλέψει. Υποχρεωθήκαμε να περικόψουμε τους μισθούς μας. Ε, οι μισθοί των ε, καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ε, περικόπηκαν κατά 30%, των τοπικών καθηγητών κατά περίπου 20%, και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε δυσκολίες πρόσληψης ε, ε, καθηγητών δευτεροβάθμιας ε, εκπαιδεύσης ακόμη και τοπικά διότι ο ανταγωνισμός μεταξύ καθηγητών επιστημών οποιαδήποτε και αν είναι η γλώσσα είναι πολύ ψηλό αυτή τη στιγμή. Υποχρεωθήκαμε να εξορθολογήσουμε όχι λόγω της έκθεσης του κ. Καβαντά αλλά λόγω της οικονομικής κατάστασης υποχρεωθήκαμε να αναθεωρήσουμε τους κανόνες ε, για το μέγεθος των τάξεων, για τον τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων. Παρά λοιπόν την αύξηση των μαθητών, ε, επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι ο προπολογισμό μας έμεινε περίπου ίδιος στα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το κόστος αναμαθητή έχει μειωθεί, μειώνεται ετησίως και προβλέπεται ίδια τάση μέχρι το 2015. Ε, ενώ ο αριθμό των μαθητών ε, αυξάνεται. Η συμβολή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μειώνεται όλο και περισσότερο αναμαθητή, διότι έχουμε περισσότερους ε, μαθητές κατηγορίας 1 και έτσι η συμμετοχή της Κομισιόν και φυσικά δεν κατηγορώ εδώ την Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο είναι εκείνα που οδήγησαν σε περικοπές και που έδωσαν σαφείς οδηγίες για το πώς να αντιμετωπίσουμε το θέμα του προπολογισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων οι μαθητές, ε, η υποστήριξη των μαθητών, όπως είπε, υπόθηκε εδώ, υπόθηκε ότι δεν προσέχουμε τους μαθητές με δικές ανάγκες. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο. Πέρυσι αναθεωρήσαμε την πολιτική υποστήριξη. Αυξάνεται ο ρυθμός ε, μαθητών με δικές ανάγκες στα σχολεία μας και αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν 800 τέτοιους μαθητές και όλοι οι τύποι παιδιομήδικες ανάγκες ενσωματώνονται τώρα. Ο ειδικό ε, προπολογισμό γι' αυτό ε, αυξάνεται παρά τη μείωση του προπολογισμού. ρημνούμε λοιπόν γι' αυτό. Εξακολουθεί να αληθεύει ότι το ποσοστό των ε, μαθητών με ειδικές ανάγκες που είναι το 3,2% αυτή τη στιγμή δεν φτάνει στο εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό αλλά αν δείτε τους αριθμούς ε, ήταν 2,7 το 2010 περίπου και τώρα έχουμε, το έχουμε αυξήσει το 3,2% συνεπώς σημειώνεται αύξηση. Πολλές συζητήσει ε, έλαβαν χώρα για τον καταμερισμό του κόστου στο cost sharing μετά από τέσσερα χρόνια πολύ δύσκολο διαπραγματεύσεων. Πέρυσι το φθινόπωρο καταφέραμε να καταλήξουμε συμβιβαστική λύση για το cost sharing Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα αυτού του κοσέρινγκ διαθέσιμα, αλλά τώρα έχει συμφωνηθεί μεταξύ όλων των κρατών μελών και των 28 ότι ο στόχος ε, για κάθε χώρα βασίζεται στον αριθμό μαθητών ανά εθνικότητα. Όπως αναφέρθηκε λοιπόν εδώ, Εάν οι χώρες ε, δεν ε, φτάνουν στο επίπεδο στόχο, μπορούν να ε, αντισταθμίσουν αυτή την έλλειψη στέλνοντας χρήματα. Αυτά τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντισταθμίσουν το κόστος μιας χώρας που στέλνει υπερβολικά πολλούς διδάσκοντες που είναι δύσκολο να βρεθούν στην τοπική αγορά διδασκόντων, για παράδειγμα, αγγλόφωνοι καθηγητές χημίας επειδή κάποια κράτη-μέλη βρίσκονται αρκετά μακριά από το στόχο, συμφωνήθηκε όλες οι χώρες από το 2015 να αυξήσουν τη συμβολή τους με 20% το έτος, κατά 20% το έτος ως το 2020, το cost sharing, ο καταμερισμός του κόστους να είναι δίκαιος και να λειτουργεί σωστά. Το Ανώτατο Συμβούλιο τον επόμενο Δεκέμβριο θα είναι το πρώτο Ανώτατο Συμβούλιο όπου πραγματικά θα εμπλακούμε σε αυτό το ζήτημα του cost sharing. Έχουν ληφθεί λοιπόν τα ζωτικά μέτρα, τα σημαντικά μέτρα, αλλά δεν έχουμε ακόμα όλη τη βοήθεια που χρειαζόμαστε στο πλευρό μας. Φέτος έχουμε 165, 67 κενές θέσεις ε, καθηγητών στο σύστημά μας. Επίσης έχουμε αλλάξει τον τρόπο δημιουργίας των θέσεων Παρατηρούμε τώρα ότι τα κράτη-μέλη, τώρα μιλάμε για το προσωπικό προσωπικό, ε, ε, υπάρχει μειωμένη βούληση αποστολή καθηγητών. Να σα το πω διαφορετικά. Είναι απολύτω ζωτικό στα ευρωπαϊκά σχολεία να διδάσκεται η μητρική γλώσσα με ανθρώπου για του οποίου η γλώσσα αυτή είναι μητρική, χωρί καμία εξαίρεση αλλά υπάρχουν κάποια μαθήματα όπως η ιστορία, η γεωγραφία, οι καλές τέχνες, ε, η γυμναστική μπορούν να διδαχθούν από ανθρώπους που δεν έχουν τη συγκεκριμένη γλώσσα ως μητρική τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις και τα μαθηματικά και οι ξένες γλώσσες σε επίπεδο 2-3-4 μπορούν να διδαχθούν από άτομα που είναι σχεδόν ε, γνωρίζουν τις γλώσσες αυτές ε, σχεδόν ως μητρική τους. Ελπίζουμε λοιπόν θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση για τα διορθωτικό μας πρόβλημα που σχετίζεται με το μεγάλο αριθμό νέων κρατών μελών που δεν αποσπούν ακόμη επαρκή αριθμό διδασκόντων. Και έτσι οι αντίστοιχοι μαθητές αυτών των χωρών αναγκάζονται να ε, φοιτήσουν στο αγγλόφωνο, στο γαλλόφωνο τμήμα. Ο κ. Καβεδάλη λέει ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τα διδακτρά. Έχει γίνει αυτό, αλλά ίσω όχι όπω αναμενόταν το Ανώτο Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα διδακτρά για του ε, μαθητέ κατηγορία 3. Αυτή είναι μια πολύ πρόσφατη απόφαση και τη σε ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου του 2013. Τέθηκε ισχύει το 2013. Αναφέρεται ότι χρειάζονται νέα τμήματα γλωσσών. Ε, πολύ προσφατά ανοίξαμε το βουλγαρικό και το ρουμάνικο τμήμα και αυτή τη στιγμή ε, συνάντησα πριν λίγο σε εβδομάδες στην εστονική αντιπροσωπεία. Ε, σχεδιάζουμε να ανοίξουμε σλοβακικό, εστονικό και λετονικό τμήμα στο εγγύς μέλλον στις Βρυξέλλες. Τώρα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην έκθεση του κ. Καβαντά υπάρχει μια σειρά στοιχείων που αφορούν τις ε, πτυχές τη παιδείας. Τη διαβάσαμε πολύ προσεκτικά Πιστεύω ότι πολλέ λάθο ε, κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Το Συμβουλίο έχει λάβει πολλέ αποφάσει βάσει των συστάσεων τη ομάδα εργασία ε, οργάνωση τη δευτεροβαθμία εκπαίδευση. Για παράδειγμα, αποφασίσαμε να ξεκινά η τρίτη γλώσσα στην πρώτη τάξη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αντί δεύτερη. Είναι θετικό. Αρχίσαμε να έχουμε προαιρετικό μαθήμα το ICT στο ετο 3 που δεν υπήρχε προηγουμένως. Θεωρούμε ότι είναι θετικό. Αποφασίσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα όπω για παράδειγμα καλές τέχνες και μουσική στο έτος 3 θα είναι υποχρεωτικά διότι θέλουμε να παρέχουμε πλήρη εκπαίδευση στους μαθητέ μα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο κόστος δεν αποτέλεσε το βασικό συντελεστή για τέτοιες αποφάσεις. Για τα υπόλοιπα, το Αρνότο Συμβούλιο αποφάσισε ότι όπως προτείνει η ομάδα εργασία πρέπει να διεξαχθεί μια εκτίμηση επιπτώσεων των άλλων προτάσεων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια μόνιμη επιτροπή, μια οργανωτική επιτροπή γιατί θα ξεκινήσει μια πρόσκληση για υποβολή προσφορών μέσα στους επόμενους μήνες. Ελπίζουμε ότι κάποια αρμόδιος οργανισμός ε, ε, ικανός για τέτοιες μελέτες. Πέρι τελευταία φορά χρησιμοποιήσαμε το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Ε, μια ομάδα του Πανεπιστήμιου του Κέμπριτζ μελέτησε τι επιπτώσει τη μεταρρύθμιση του Μπακαλωρέα πριν αυτέ τεθούν σε ίσχυ. Ζητάμε αυτή τη στιγμή κάτι παρόμοιο. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα ποιο οργανισμό ή ποιο πανεπιστήμιο θα μπορούσε να διεξάγει τη μελέτη. Αλλά η πρόσκληση για υποβολή προσφορών θα ξεκινήσει. Δεν προσεγγίζουμε λοιπόν τα θέματα μόνο από την οικονομική άψη. Πραγματικά με μεγάλη προσοχή προσπαθούμε να διατηρήσουμε ό,τι καλό υπάρχει για το Ευρωπαϊκό Μπακαλόρεα. Δεν έχω κάποια διαφάνεια για το Ευρωπαϊκό Μπακαλόρεα, αλλά μπορώ να σας πω ότι εκτιμάται ιδιαίτερα από τα πανεπιστήμια. Να ενημερώσω την κυρία Χόνιβαλ ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας στην ιστοσελίδα των σχολείων μας και στο Υπουργείο Παιδείας μας που δείχνει πώς ε, υψηλό ποσοστό επιτυχών των έχουν τα σχολεία μας στα Βρετανικά πανεπιστήμια. Μεγάλο ποσοστό σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερε δυσκολίες οι μαθητές μας να λάβουν καλές προσφορές από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Θα έλεγα λοιπόν ότι η αξία του Ευρωπαϊκού Μπακαλωρέα υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει. Το ίδιο ισχύει και για τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ολλανδικά πανεπιστήμια ακόμη και σε πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης. Δεν έχω όλες τις λεπτομέρειες, ε, αλλά ένα σημείο που αναφερθώ στο τέλος του γράφου ε, αφορούσε ε, τις επαναλήψεις τους, δηλαδή τις αποτυχίες. Πράγματι θεωρείται ότι είχαμε υψηλό ποσοστό αποτυχόντων. Ε, υιοθετήσαμε 19 μέτρα το 2010 για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό. Το παρακολουθούμε στενά και είχαμε αρκετά καλά αποτελέσματα. Από το ποσοστό 2007 2010, 2,7 έχουμε φτάσει σήμερα στο 1,2. ατόμων που χρειάστηκε να επαναλάβουν τις τάξεις. Δεν συμμερίζομαι λοιπόν την απεσιοδοξία σας. Τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι... Έχουμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν στι Φρυξέλλες, στο Μόναχο, στη Φραγκφούρτη. Σε πολλά μέρη έχουμε υπερβολικά πολλούς μαθητές που επιθυμούν ε, να πάνε σε σχολεία αυτά και να φοιτήσουν τα σχολεία αυτά και δεν έχουμε αρκετό χώρο. Είναι πραγματικά κρίμα. Η καταστάση στο Λουξεμβούργο είναι πολύ εντάξει. Υπάρχει ένα νέο σχολείο με πολλούς περισσότερους μαθητές κατηγορίας 3. Αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου να επεκτείνουμε ακόμα και αυτό το σχολείο στο μέλλον. Στο Ανώτο Συμβούλιο έχουμε αποφασίσει πολλά μέτρα σε δύσκολε εποχέ για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Τα σχολεία μα είναι πιο δημοφιλή από ποτέ. Έχουμε ένα πρόβλημα υπερβολικά υψηλού αριθμού μαθητών. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Τα διαπιστευμένα ευρωπαϊκά σχολεία και το νέο σύστημα αυτό, όλα αυτά πάνε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Τουλάχιστον σε σχέση με το follow από τη συνέχεια, σε σχέση με την έκθεση αυτή που ελήφθη σοβαρά υπόψη στις ε, παρατηρήσεις, σε σχέση και με τα όσα γίνονται. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να ακούσουμε εκείνους που μας προσεγγίζουν διαρκώς και έχουν παράπονα και παραπονούνται δεν είναι όλα τα παράπονα που έχουν τώρα αξιολογηθεί και διευθετηθεί από τον Γενικό Γραμματέα ή από τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ανώτατου Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο ε, ε, από πλευράς Inter Άραντ. Ε, είχαμε και την ε, εκλογή πρόσφατα. Ναι, Πρόεδρε, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την προσωπική σας ε, μέρημνα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά σχολεία και ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε για να υπάρξει ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις. Κόρνης Μπάρβα είναι το όνομά μου και έχθες από χθε το απόγευμα έχω εκλεγεί Πρόεδρος αυτού του σώματος που όπως γνωρίζετε συντονίζει και εκπροσωπεί τις ενώσεις και συλλόγους γονέων στα ευρωπαϊκά σχολεία. Οι Interparents συμμετείχαν στη στρογγυλή τράπεζα του κ. Καβαντά και ενημέρωναν αυτή την Επιτροπή σε τακτά διαστήματα για τη συνέχεια ή έλλειψη συνέχειας και παρακολούθησης που είχε παρατηρηθεί. Θεωρούμε ότι είναι σοβαρά προβλήματα αυτά τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τα ευρωπαϊκά σχολεία και αυτά ανοιχνεύθηκαν σε σχέση με το 2002 ήδη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε σχέση με την επίλυση τους για να υπάρξει ένα πιο ισοδίκαιο, ένας πιο δίκαιος τρόπος επιμερισμού των, ε, ε, του κόστους και των δαπανών. Τόσο σοβαρά είναι αυτά τα προβλήματα που ε, το Συμβούλιο για την ε, Νεολαία και την Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό συζήτησε το θέμα και είχαμε και μια έκτακτη συνεδρίαση που ζητήθηκε να ε, συγκληθεί των Υπουργών Παιδείας και Εκπαίδευσης ώστε να συζητηθούν τα θέματα της πρόσφατης κρίσης. Θα λέγαμε τώρα μια τέτοια σύγκληση, μια τέτοια συνεδρίασης έχει κατεπήγοντα χαρακτήρα παρότι ακούμε μήνες μετά κάποια πράγματα δεν υπάρχει αξιόπιστη λύση ενώπιόν μας. Και η μεγάλη ζήτηση Γάλλων, Γερμανών και άλλων καθηγητών και Άγγλων είναι απορρέει από το ότι σε αυτές τις τρεις γλώσσες διδάσκονται είτε ως πρώτη, δεύτερη, τρίτη γλώσσα οι μαθητές στα ευρωπαϊκά σχολεία. Και πρέπει να δούμε ότι δεν είναι δυνατόν το κόστος ε, να επιμερίζεται με αυτόν τον τρόπο και το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είχε οξύτατα αποτελέσματα και πολιτικά και επιτόπου στα σχολεία. Απουσιάζουν λοιπόν καθηγητές ε, στο σύστημα συνολικά και είναι σημαντική αυτή η απουσία. Και η επικεφαλής ε, σε σχέση με τα όσα έχουν συμφωνηθεί από πλευρά των κρατών μελών δεν υπάρχει όμως μηχανισμός που να έχει συμφωνηθεί για την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και με το καλύτερο ακόμα σενάριο ο αριθμός των καθηγητών αυτών είναι αξιοπερίεργα χαμηλότερος από έτος σε έτος. Ποτέ δεν διασφαλίζονται αυτοί οι καθηγητές έγκαιρα και ούτε μέχρι και το Σεπτέμβριο και έχουμε και το 20% αύξησης ε, που μέχρι το 2020 με τις προοπτικές που υπάρχουν δεν θα υπάρχουν καθηγητές διαθέσιμοι. Και οι υποσχέσει να υπάρξουν, θα υπάρξουν εναλλακτικέ δυνατότητες χρηματοδότησης είναι γενικόλογε και αφηρημένε και μετέωρε Και όλα αυτά παρότι αυξάνεται ο γενικό πληθυσμό των μαθητών, ο αριθμό των μαθητών. Και υπάρχουν αισιόδοξε υποθέσει ότι πρώτον κάποιε χώρε θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν εθελοντικά σε ένα εθελοντικό πλαίσιο Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία ή Ολλανδία, καθώ επίση και το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη δομή. Δεύτερον, υπόθεση ότι η αγορά χωρίς περιορισμό θα μπορεί να διαθέτει τέτοιου είδους καθηγητές στα αναγκαία μαθήματα. Τρίτον, η συνέχεια στην διδασκαλία μπορεί λέει να διασφαλιστεί με αυτού του είδους τους καθηγητές που όμως έχουν συμβάσεις περιορισμένου χρόνου περιορισμένης απασχόληση Είναι λοιπόν πολύ απογοητευτική η συνολική εικόνα, αλλά δεν είναι μόνο η εκπαίδευση των παιδιών τη μελλοντική γενεά που διακυβεύεται, είναι και η μοναδική αυτή προσέγγιση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά σχολεία, την εκπαίδευση και το ευρωπαϊκό απολυτήριο. Είναι ένα πρότυπο που όλο και περισσότερο ακού, ακούμε ότι τα κράτη-μέλη υιοθετούν στη Φινλανδία, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία και θα συμφωνούσαμε ότι αυτή η επέκταση είναι μάρτυρας ε, κατά μαρτυρή ότι το όραμα εκείνο μιας ευρύτερης ε, προσέγγισης, ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής προσέγγισης μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας με ρίζες στον ίδιο τον πολιτισμό του κάθε μαθητή θα είναι στερεά θεμέλια και θα υπάρχει μια δυνατότητα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και είναι και μια πρόκληση. Αυτή η συζήτηση λοιπόν για τα ευρωπαϊκά σχολεία πρέπει να αποτελέσει άρρηκτα μέρος της συζήτηση, ως τμήμα της συζήτησης για το τι θα γίνει σε σχέση με την εκπαίδευση γενικότερα και το θέμα της, του συμμερισμού, του επιμερισμού του κόστους. Ευρύτερη συζήτηση έγινε σε σχέση με μελέτες για το πώς πρέπει να χρηματοδοτούνται αυτά τα σχόλια. Ριζοσπαστικές ε, προτάσεις, ριζοσπαστικές αλλαγές σε αυτές τις προτάσεις θα μπορούσαν να μεταβάλουν σε πολύ ε, σημαντικό βαθμό ακόμα και τη δομή ε, του, των μαθητών σε αυτά τα σχολεία και βλέπουμε ότι δεν ήταν αυτό εκείνο το οποίο στόχευε να επιτύχει, να επιτευχθεί ο κύριος Καβαντά. Χαίρομαι όμως ε, για το ότι ακούγεται ότι τουλάχιστον κάποιες από αυτές τις προτάσεις ε, θα υποβληθούν σε μια εξωτερική αξιολόγηση ως διαδικασία. Αναμένουμε και προσδοκούμε να δούμε τι θα γίνει με κομμένη την ανάσα. Κάποιες προτάσεις ε, που επιτείνουν το πρόβλημα του κόστους και των δαπανών και στις τρεις κυριότερες γλώσσες και μάλιστα επιζήμιο είναι αυτό για τις αναγκαιότητες της πολυγλωσσικής κατάρτισης ενός πολυγλωσσικού καθεστώτος. Και να μην ξεχνάμε και την ενδυνάμωση της εθνικής ταυτότητας, πολιτισμικής, πολιτιστικής ταυτότητας των παιδιών, των μαθητών, που έχει και αυτή σημαντική διάσταση. Και δεν είναι μόνο το θέμα της κατανόησης της γλώσσας ή των εκφράσεων μιας γλώσσας. Είναι το θέμα ότι οι καθηγητές πρέπει να κατανοούν το εθνικό σύστημα από το οποίο προέρχονται οι μαθητές στα ευρωπαϊκά σχολεία και στο οποίο θα επιστρέψουν μετά τις ε, σπουδές τους σε ένα τέτοιο σχολείο όταν επιστρέψουν στη χώρα τους. Δεν είναι κάτι το οποίο σύντομα βραχυπρόθεσμα μπορεί να παρασχεθεί, πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα συνοδεύει μακροπρόθεσμα όλη την εκπαίδευση στα ευρωπαϊκά σχολεία. Γιατί καμιά φορά, αν δεν τα προσέξουμε αυτά, μπορεί να χαθεί, να απολεστεί. Σε σχέση τώρα με τα αναφέρει ο κύριος Καβαδά, για τις ε, ανάγκες για τη χρηματοδότηση και τις συστάσεις που υποβάλλονται για το 2011 στο ψήφισμα του Ευρω... της Ευρωβουλής λυπούμαστε που επανερχόμαστε σε εσά και δεν έχουμε καλύτερα μαντάτα να σας γνωστοποιήσουμε, να σας ε, δώσουμε. Αν θέλει κανείς να το πιστέψει κάτι τέτοιο, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, τα πράγματα κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, ω συνήθως συζητούνται κτλ. Βλέπουμε όμως τις επιπτώσεις ποιες είναι στα σχολεία. Ο αριθμός των μαθητών, ακούσαμε επανειλημμένα, αυξάνεται διαρκώς. Έχουμε και μάλιστα υψηλότερα δίδακτρα τα οποία απαιτούνται. Έχουμε συρρυκνωμένους ε, με περικοπές προϋπολογισμούς. Τα θέματα ασφάλειας έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη του, Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλο και λιγότερη έμφαση δίνεται στις, ε, στη μητρική γλώσσα. Κλείνουν και ε, γλωσσική κλάδη όταν δεν υπάρχει, ας το πω υποστήριξή τους. Ε, έχουμε και περιορισμό των ορών και πάλι εδώ έχουμε το θέμα των στελεχών, των καθηγητών που απουσιάζουν, λείπουν και βλέπουμε ότι από πλευράς ε, της εθνικής συνιστώσας πρέπει να μπορεί να διασφαλίζεται ο αριθμός των αναγκαίων καθηγητών. Βλέπουμε ότι συρρυκνώνεται όμως. Θα πρέπει λοιπόν ε, ο διακυβερνητικός ρόλος των ευρωπαϊκών σχολείων να ενδυναμώνεται και όχι να αποδυναμώνεται μέσα από όλα αυτά. Ε, χρειάζεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο μεγαλύτερη προσπάθεια. Μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί μια αηφορία στις λύσεις που θα δοθούν για τα ευρωπαϊκά σχολεία. Στις προηγούμενες ε, προσπάθειες που καταβάλατε και ε, σε σχέση με την εκπροσώπηση των γονέων, με το, την έντονη δουλειά που έχουμε κάνει, η εντύπωση μας είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να είναι κανείς αισιόδοξο και να υιοθετεί μια επικοδομητική προσέγγιση. Υπάρχει απογοήτευση, χρειάζεται όμω ένα πιο μακροπρόθεσμο όραμα ως συνιστόσα και χρειαζόμαστε καθηγητές ήδη το Σεπτέμβριο διαθέσιμους. Να μην το ξεχνάμε ότι έχουμε μια γενεά μαθητών τώρα, σήμερα που χρειάζονται να καλυφθούν οι ανάγκες τους εκπαιδευτικά σήμερα. Ευχαριστώ. I still have a... Ναι, έχω, πάλι, έχω ακόμα μια ερώτηση από την έκθεση του Ζεράρ Περί, ήδη από την εποχή εκείνη πριν από αρκετό καιρό. Εκείνη την εποχή είχαμε θέσει το εξή θέμα. Πολλοί από τα, τους μαθητές που τελικά δεν φτάνουν στο μπακαλωριά αλλά διακόπτουν νωρίτερα το σχολείο και χωρίς ε, απολυτήριο. Είχαμε θέσει το εξή ερώτημα. Είναι δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι μπορεί να υπάρξει μεσοπρόθεσμα μια διακοπή του σχολείου. Έχει ζητηθεί κάτι σχετικά στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου. Ε, α, στα γερμανικά το λένε Mittlere Reife. Είναι ένα είδος απολυτηρίου ε, για τα παιδιά εκείνα τα οποία δεν φτάνουν στο μπακαλωρεά. Ε, δεν ξέρω αν προβλέπετε μια τέτοια δυνατότητα ή αν έχει συζητηθεί σχετικά το θέμα αυτό στο Ανώτατο Συμβούλιο. Κύριος Κίβινεν, ε, πράγματι το θέμα αυτό ε, σε σχέση με τις εξελίξεις στις χώρες μέλη. Σε όλο και περισσότερες χώρες στην Ευρώπη υπάρχει ένα είδος σχολικού διπλώματος στην ηλικία των 15-16 ετών και έτσι ε, παιδιά που επιλέγουν να πάνε σε τεχνικά σχολεία ή να ακολουθήσουν μια επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να επιλέξουν μεταξύ αυτών των εναλλακτικών δυνατήτων. Στην ευρωπαϊκά, στα ευρωπαϊκά σχολεία ε, έχουμε μόνον τον μπακαλωριά. Τώρα, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της ομάδας εργασίας για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στο πλαίσιο της ομάδας αξιολόγηση, ότι είναι αναγκαίο για τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο να έχουν κάποιο είδος ε, πιστοποίησης για τα όσα έχουν κάνει μέχρι τότε. Στο Ευρωπαϊκό Σχολείο, για παράδειγμα, ε, σπουδάζουν γλώσσες από την ηλικία των 6 ετών, ε, συνήθως με καθηγητές που είναι αυτή η γλώσσα μητρική τους και πραγματικά εκπαιδεύονται πολύ καλά. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια ομάδα αξιολόγησης που να πιστοποιεί αυτές τις ικανότητες των μαθητών που διακόπτουν το σχολείο, ούτω ώστε να υπάρχει δυνατότητα για όλους μας τους ε, μαθητές, ναι μεν να μπορούν να συνεχίσουν μέχρι τον μπακαλωρεά, αλλά αυτοί οι οποίοι θέλουν να στραφούν αλλού να μπορούν να έχουν μια αναγνώριση αυτών που έχουν μάθει μέχρι τότε ή του επίπεδου, να πιστοποιείται το επίπεδό τους ε, για τα μαθήματα αυτά, τις γλώσσες παραδείγματι. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Έχω άλλη μια ερώτηση. Ε, συχνά μου λένε ε, ότι αυτοί οι οποίοι είναι κάτοχοι μπακαλωρεά, ευρωπαϊκού μπακαλωρεά, στη Γερμανία, εφόσον δεν μεταφράζεται, δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν. Δεν ξέρω, ε, υπάρχει μόνο σε μία γλώσσα ή είναι δυνατόν να υπάρξει σε πολλές μεταφράσεις ούτω ώστε οι υπηρεσίες των αντίστοιχων χωρών να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, να το αξιοποιήσουν μάλλον. Ε, δεν ξέρω, ήθελα να μου πείτε κατά πόσο έχετε και εσείς γνώση του σχετικού προβλήματος. Καταρχήν, για τους μαθητές που εγκαταλείπουν το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων ε, σε 28 χώρες μέλη ε, θα υπάρξει ένας ε, πίνακας αντιστοιχίας των μαθημάτων στα ευρωπαϊκά σχολεία, αντιστοίχησης με τα μαθήματα στα, στις διάφορες χώρες μέλη. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά ε, στις χώρες που έγιναν ε, πρόσφατα χωρίς μέλη δεν υπάρχουν ε, ειδικέ ε, γνώσεις για αυτά τα θέματα. Τώρα, όσον αφορά τον μπακαλωρεά, αυτό γίνεται στο αντίστοιχο γλωσσικό τμήμα. Το επόμενο καλοκαίρι θα βάλουμε και τα βουλγαρικά, τα ρουμανικά, γλώσσες που ήταν αδύνατον να διδαχθούν στο πλαίσιο του παλαιού συστήματος. Τώρα λοιπόν θα δίδουμε το μπακαλωρεά σε όλες αυτές τις γλώσσες. Ε, μάλιστα. Συνάδελφοι, ποιος θέλει να λάβει τον λόγο τώρα. Κύριε Τάκουλα, παρακαλώ. Κοίταξε που Σας ευχαριστώ πολύ. valaisevaa, tiedetään missä mennään, mutta... Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ για μια διεξοδική ε, παρουσίαση που μας κάνει να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε ως μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Και πρακτικά, επειδή τα ευρωπαϊκά σχολεία είναι πρωτοπόρα ιδρύματα, ήταν πρωτοπόροι και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνο ήπιες εξουσίες, soft powers, δυνατότητες συντονιστικές όσον αφορά την εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν με τον καλύτερο τρόπο να προαθούν από αυτές τις κοινότητες τα θέματα των ευρωπαϊκών σχολείων. Είναι κάτι που εμπλουτίζει πολύ τη ζωή μας ε, και, την, ε, και είναι πολύ διαφωτιστικό. Όμως αυτό που μας ανησυχούν είναι ότι αυτά τα θέματα που αφορούν τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ευρωπαϊκά σχολεία, για παράδειγμα στο Βέλγιο, όπου γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα καθηγητών, για παράδειγμα, Η όρια απασχόλησή του στι συμβάσει πρέπει να είναι συντονι... Ε, και μας ανησυχεί το θέμα της διαθεσιμότητας των καθηγητών. Φαίνεται ότι είναι μεγάλη η δυσκολία να εξευρεθούν τα αναγκαία στελέχη, να στελεχωθούν τα σχολεία όπως πρέπει. Και ένα άλλο θέμα, εδώ η παιδεία, η εκπαίδευση είναι ο τομέας εκείνος που υφίσταται τα μάλα από μια τέτοια κατάσταση. Και βλέπουμε ότι σε σχέση με τα περισσότερα μαθήματα, τα γλωσσικά μαθήματα, στα γερμανικά ή στα γαλλικά, φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα να στελεχωθούν ε, τα σχολεία με τον αναγκαίο αριθμό κατάλληλα εκπαιδευμένων και ε, με τις ικανότητες που απαιτείται καθηγητών και χρειάζονται εδώ και οι ε, ε, δυνατότητες αναφοράς και ε, προσαρμογής στον εκπαιδευτικό τομέα και τις ανάγκες του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει και ανησυχούμε. Και τα θέματα τα κτηριακά ή των εγκαταστάσεων αναφέρθηκαν. Απουσία υποδομών, σχολείων, κτηρίων κτλ. Βλέπουμε όμως ότι πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές σε σχέση με τα ευρωπαϊκά σχολεία ώστε σε σχέση με τους, ε, τις ε, επισκέψεις ε, που κάναμε δεν δίνουν καθόλου την εντύπωση ελιτιστικών σχολείων. Δεν είναι ελιτιστικά σχολεία, πρέπει όμως να υπάρχει η δυνατότητα να έχουν τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες να επιτύχει το έργο τους και όσοι πάνε σε αυτά τα σχολεία, όσοι στέλνουν τα παιδιά τους σε αυτά τα σχολεία να έχουν μια προοπτική, τα παιδιά αυτά να εκπαιδευτούν, να κατατιστούν κατάλληλα όπως πρέπει και να έχουν τη δυνατότητα με τον πιο επαρκή τρόπο να καλύψουν τις ανάγκες τους σε σχέση με τους ε, καθηγητές για παράδειγμα και τον αριθμό τους που υπάρχει πρόβλημα εκεί. Η υπερβολική συγκέντρωση μαθητών σε κτίρια που δεν επαρκούν, εξωτερικά ζητήματα όπως ασφάλεια, θέματα ασφάλειας, όλα αυτά υπονομεύουν τη γενική, ας το πω έτσι, εικόνα αυτών των σχολείων ή το πώς παρουσιάζονται αυτά τα σχολεία στους πολίτες. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθούν αυτά τα πράγματα και είναι δουλειά μας εμείς στα κράτη-μέλη να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότησή τους θα βαίνει καλώς και δεν θα υπάρχουν προβλήματα λόγω των πολιτισμικών διαστάσεων που έχουν αυτά τα θέματα. Δεν είναι δικό μας ε, το έργο αυτό δυστυχώς, είναι έργο των κρατών μελών. Εμείς δεν μπορούμε να αναμειχθούμε με κανένα τρόπο, μπορούμε μόνο προτάσεις να υποβάλουμε και αυτές πρέπει να τύχουν συνέχεια. Εσείς παρακολουθείτε. Έχω μια ιδιαίτερη ερώτηση. Αναφέρατε τις Βρυξέλλες. Ε, δεν ξέρω, έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο από τα διορθωτικά ταμεία στην ενότητα της, ποιότητα, της ισότητας, κατά πώς θα μπορούσε να υπήρχε κάποια δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε ένα κτίρια για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα των κτίριων. Το Ανωτό Συμβούλιο έχει υπογράψει μια συνθήκη με το Βέλγιο το βελγικό κράτος έχει την υποχρέωση να μας παράχει τα κτίρια. Είναι πολύ δύσκολο για μας να αιτιολογήσουμε οποιαδήποτε δαπάνη για κτίρια, διότι υπάρχει αυτή η σύνθηκη. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τέτοια δαπάνη για οποιοδήποτε άλλο κονδύλιο του προπολογισμού. Συνεπώς ε, θα εξαρτηθεί το όλο ζήτημα από το Βέλγιο, από τη φιλοξενούσα χώρα, τη χώρα υποδοχής. Να σας πω δύο λόγια παραπάνω για την κατάσταση τη Βρυξέλλες, όπως έχει μέχρι στιγμές πρόεδρος των γονέων, του Συλλόγου Γονέων είναι χαρούμενος διότι είναι γονέας ε, για παιδιά πάνε σε ένα σχολείο που έχει εξαιρετικές ε, εγκαταστάσεις. Το Λάκεν μπορείτε να το επισκεφθείτε. Είναι ένα καταπληκτικό κτίριο σύμφωνα με όλα τα πρότυπα. Εκεί έχουμε ακόμα 800 ελεύθερες θέσεις μαθητών. Από την άλλη όμως ε, Έχουμε τους μαθητές μας από το σχολείο του Ουκλε σε κτίρια του Μπέρκενταλ και 400 θέσεις περίπου με αναχρησιμοποιητές. Τη φετινή σχολική χρονιά λοιπόν έχουμε θέσεις. Το πρόβλημα είναι ότι το Ανώτο Συμβούλιο ε, εγγυήθηκε στους γονείς ότι δεν θα μετακινηθεί κανένας μαθητής από το ένα σχολείο στο άλλο. Και εμείς τηρούμε αυτή τη δέσμευση. Δεν μπορούμε λοιπόν να πάρουμε μαθητές από ένα σχολείο με υπερβολικά πολλούς μαθητές για να τους πάμε σε ένα άλλο. Ε, συνεπώς γεμίζουμε τις νέες θέσεις με τους νέους μαθητές για να σας δώσω τα πιο τελευταία νέα που έλαβα μέσω email. Έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη φάση εγγραφών για τον επόμενο Σεπτεμβρίο εδώ στις Βρυξέλλες και έχουμε ένα νέο ρεκόρ 1600 εγγραφών ήδη μέχρι στιγμή 750 εγγραφέ αντιστοιχούν σε παιδιά νηπιαγωγείου και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετού χώρου νηπιαγωγείου, όλα είναι γεμάτα. Υπάρχει λοιπόν μια δημογραφική μεταβολή στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την οποία δεν ήταν έτοιμα τα κτίρια μα. Με τα νέα κράτη-μέλη πριν από 8-9 χρόνια ήρθαν πολλοί νέοι υπάλληλοι νέα ηλικία με 5-6 χρόνια εμπειρία οι οποίοι παντρεύτηκαν και έχουν μικρά παιδιά. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτή τη οικογένειακή κατάσταση στα σχολεία μας. Εμείς ε, υπολογίζουμε ότι οι χώροι το, για τα νηπιαγωγεία μας ε, θα πρέπει να επεκταθούν. Υπάρχουν υψηλές ανάγκες. Έχουμε λοιπόν κάποιο αχρησιμοποιητό χώρο αυτή τη στιγμή. Αλλά η κατάσταση στα σχολεία είναι δύσκολη. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Δώσαμε δυνατότητα στους 3.500 μαθητές του σχολείου του Βολιβέ για να πάνε σε άλλο σχολείο και μόνο 8 εκδήλωσαν τέτοια επιθυμία. Είναι πολύ αγαπητό το σχολείο του Βολιβέ. Και έχει δοθεί και αυτή η υπόσχεση από το Νότο Συμβούλιο ότι δεν θα μετακινηθούν μαθητέ. Συνεπώ, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γεμίσουμε τον κοινό χώρο με του νέου μαθητέ. Κυρία Κώστα, πεις. Η κυρία Κώστα, παρακαλώ, ευχαριστώ. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Και η περιγραφή που ακούσαμε από τους διαφόρους, ε, όπως κατάλαβα, υπάρχει κάποια προσπάθεια προσαρμογής ε, βάσει των κατευθύνσεων που έχει δώσει το Κοινοβούλιο. Φυσικά το θέμα της χρηματοδότησης δεν έχει πληθεί και αποτελεί ακόμα το επίκεντρο και αυτό φυσικά δεν διευκολύνεται από το γεγονό ότι είναι εθελοντική συμμετοχή από τα κράτη-μέλη, ειδικά αυτέ τι εποχέ κρίση, ε, όπου πληθεί και την Ιταλία, για παράδειγμα. Δεν έχουμε χρήματα να χρηματοδοτήσουμε τα δικά μα σχολεία καλά-καλά. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Βάσει ποια βάση μιλάμε για τα νέα σχολεία που θέλουν να ανοίξουν σε διάφορε χώρε, άκουσα τα Λίν, Μπρίντεζι και άλλε ευρωπαϊκέ πόλει. Θέλω να με εξηγήσετε, όσον αφορά τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνονται δεκτά τα νέα αιτήματα, πέραν της δέσμευσης των κρατών μελών. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα κριτήρια βάσει των οποίων αποφασίζεται ένα σχολείο αντί για κάποιο άλλο. Και ποια είναι η διαδικασία λήψη απόφαση για ε, το άνοιγμα των σχολείων αυτών και με ποιο τρόπο συμμετέχει το Ανατό σε αυτή τη συζήτηση. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ περισσότερα είναι τα σχολεία στο βορρά τη Ευρώπη από ότι στο νότο. Και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε. Κάτι άλλο επίση. Πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα Ζητώ συγγνώμη που έχω την πλάτη μου προς τα άτομα στα οποία απευθύνομαι. Ενδιαφέρον το αποτέλεσμα μείωση των ατομών που χρειάζεται να επαναλάβουν την τάξη. Καθώς και το ζήτημα του ανοίγματο των σχολείων με παιδιά με ειδικές ανάγκες, για παιδιά με ειδικέ ανάγκες. Ήθελα να πείτε, αυτή η μείωση των αποτυχιών σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη δράση που ανέλαβε το σχολείο και τι τύπου δράση ήταν αυτή ή μήπως ε, ήδη ευθύ εξ αρχής γίνονται δεκτά άτομα υψηλότερου δηλαδή είναι αποτέλεσμα αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας των σχολείων ή είναι αποτέλεσμα υποδοχής ε, καλύτερων μαθητών, ε, μαθητών με περισσότερες δυνατότητες, ουσιαστικά ικανότητες. Είναι πολύ ενδιαφέρον το στοιχείο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να το αναλύσουμε. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστούμε τη Σίλβια. Άλλες ερωτήσεις. Γενικό Γραμματέας, παρακαλώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρησε το κανονισμό για τη δημιουργία των πιστοποιημένων ευρωπαϊκών σχολείων πέρσι και απλουστεύθηκαν και διευκρινίστηκαν στη βάση της, ε, ε, των προτάσεων των χωρών ε, μελών και μπορούν όλα αυτά να συζητηθούν στην κοινή επιτροπή όπως κάναμε σήμερα το πρωί για το πρέντιζι. και στη συνέχεια θα πρέπει κάθε χώρα να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια μπορεί να ανοίξει το σχολείο. Δεν γίνεται επιλογή, εάν θέλετε. Απλώς θέλουμε να εγγυηθούμε το υψηλό επίπεδο ποιότητας των ευρωπαϊκών σχολείων και ε, ιδιαίτερα στην ε, οργάνωση των ε, σπουδών που γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Άρα λοιπόν είμαστε ανοιχτοί για όλα τα διαπιστευμένα σχολεία. Τώρα όσον αφορά τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, καθώς και τους μαθητές που διακόπτουν το σχολείο. Εμείς δεν επιλέγουμε τους μαθητές μας. Βεβαίω υπάρχει μια φυσική επιλογή, για παράδειγμα στις Βρυξέλλες, όπως είπε ο κύριος Καβαντά, όπου, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολύ αυστηρή πολιτική εγγραφών σχεδόν όλοι 1600 μαθητές ε, για του χρόνου είναι μαθητές της κατηγορίας Α. Ίσως 52 από την κατηγορία 2 και 10 ή 11 της κατηγορίας 3. Άρα λοιπόν η επιλογή γίνεται κάπου αλλού και όχι εντός του δικού μας σχολικού συστήματος. Αλλά υπάρχουν σχολεία που έχουμε περίπου 70% μαθητές ε, από την κατηγορία 1. Υπάρχουν όμως και σχολεία όπου η κατηγορία αυτή των μαθητών 1 είναι πιο χαμηλή. Άρα λοιπόν δεν επιλέγουμε ε, τους μαθητές ε, με υψηλές ικανότητες αλλά στη βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης ε, ΠΙΣΑ ε, ελήφθη υπόψη και το, ε, εκπαιδευτικό, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Αυτό είναι ο καθοριστικός παράγων. Η Κομισιόν παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη συζήτηση. Ακούσαμε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την παρακολούθηση της έκθεσης Καβαντά και πραγματικά συμμεριζόμαστε τα βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει να παρακολουθηθούν και τα οποία επεσήμανε ήδη ο κύριος Καβαντά και που αφορούν τη χρηματοδότηση, την απόσπαση, την ε, μεταρρύθμιση της ορμάθμιας εκπαίδευσης και το πρόβλημα των υπεράριθμων μαθητών. Αρκετές απαντήσεις δόθηκαν εδώ και αναμένουμε τώρα την μεταρρύθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη σχετική αξιολόγηση. Η Κομισιόν δεν έχει τη συνήθεια να ανακατεύεται σε παιδαγωγικά θέματα, γιατί εδώ δεν έχουμε την αρμοδιότητα, αλλά το αφήνουμε στους εμπειρογνώμονες των χωρών μελών, που είναι πολύ πιο αρμόδιοι από εμά για ζητήματα εκπαιδευτικού περιεχομένου και που είναι σε θέση να κάνουν τη σύνδεση με το επίπεδο των πανεπιστημίων των χωρών μελών, ούτως ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων να μπορεί στη συνέχεια να συνδυάζεται με ε, τις ε, προϋποθέσεις όδου στα πανεπιστήμια. Τώρα όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η θέση της Επιτροπής σε σχέση με το cost sharing είναι ότι βεβαίω θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα πράγματα. Η συμφωνία ε, που απαιτεύθηκε δεν ήταν και πολύ φιλόδοξη. Η Κομισιόν είχε προβλέψει ένα πολύ γρηγορότερο phasing in και τελικά κατέληξε σε μια πιο σημαντική συμμετοχή των κρατών μελών. Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι αυτό το οποίο είναι ο κοινός, ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής που πετύχαμε και συμμετείχαμε πραγματικά σε αυτή την προσπάθεια όλοι, και τώρα περιμένουμε την εφαρμογή το 2015 και θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος. Τώρα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, θέμα εδώ αναφέραμε τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των αποσπασμένων καθηγητών και θα ήθελα να την προσοχή των Ευρωβουλευτών στο γεγονός ότι όλες οι αναθεωρήσεις των ε, προϋποθέσεων ε, των οικονομικών προποθέσεων της εργασίας των καθηγητών έγιναν σε συνάρτηση με την αρχή μιας παράλληλης ισχύω της ε, ε, του δημόσιου λειτουργήματος και των ευρωπαϊκών σχολείων από την άλλη. Και ε, λάβαμε υπόψη όλες τις προσαρμογές που έγιναν στα ευρωπαϊκά σχολεία. Όσον αφορά εν γέννη στους πόρους μας, πραγματικά θέλουμε να δηλώσουμε την εμπιστοσύνη μας στην Επιτροπή αυτή για να μας υποστηρίξει έναντι της Επιτροπής Προπολογισμού, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά σχολεία. Τώρα, όσον αφορά τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό των μαθητών στα ευρωπαϊκά σχολεία, θέμα που αναφέρθηκε σε πολλέ από τι παρεμβάσει, θα ήθελα να σα εξασφαλί... διαβεβαιώσω ότι ο κύριο Σεφκοβιτ ε, έχει σε εβδομαδιαία βάση επαφέ με τι βελγικέ αρχέ για να τις παροτρύνει να λάβουν μια σχετική απόφαση όσον αφορά την στέγαση ε, του 5ου Ευρωπαϊκού Σχολείου στις Βρυξέλλες αλλά δυστυχώς για λόγους που αναφέρθηκαν από τη βελική αντιπροσωπεία, οι προσπάθειες αυτές ε, δεν κατέληξαν σε κάποιο αποτέλεσμα, παρόλα αυτά αποτελούν προτεραιότητα για μας. Είμαι στη διάθεσή για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν δόθηκε απάντηση από τους Βέλγους σε αυτό το ερώτημα. Και γι' αυτό δεν είναι τώρα θέμα εδώ για μια υπερώτηση για παράδειγμα. γιατί στο Βέλγιο ακόμα δεν υπάρχει απάντηση που να δόθηκε. Ίσως οφείλεται στις εκλογές. Τι να πούμε. Δεν το ξέρουμε. Ίσως ένας από τους εκπροσώπους του Βελγίου θα ήθελε κάποια παρατήρηση να κάνει. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποια παρατήρηση. Δεν θέλετε να παρέμβετε. Ωραία, εντάξει. Ε, λοιπόν θα έλεγα τότε και εξ ονόματος του κυρίου Καβαντά μπορώ να μιλήσω και εξ ονόματός του εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου για τη συμμετοχή σας για τις αξιόλογες πληροφορίες που μας έδωσε ο Γενικός Γραμματέας που κατέδειξαν ότι σε κάποια σημεία σίγουρα σε σχέση με την έκθεση του Κοινοβουλίου όπως παρουσιάζεται από τον κύριο Καβαντά ακολουθείτε αυτές τις θέσεις. Ξέρουμε ότι δεν έχουν επιτευχθεί όλα όπως θα επιθυμούσαμε. Ξέρουμε ότι δεν έχουν επιληθεί ικανοποιητικά αυτά τα προβλήματα. Το κατανοούμε. Ως γονείς υπάρχουν άλλες απαιτήσει σε σχέση με το τι μπορεί να επιτευχθεί. Σε όλα τα σχολεία συμβαίνει κάτι τέτοιο, σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία συμβαίνει αυτό. Σήμερα όμως είχαμε μια συζήτηση θα έλεγα που μπόρεσε να μας δώσει ίσως μια καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει. Ελπίζουμε ότι θα δοθεί συνέχεια στις καλές συμβουλές και προτάσεις του κυρίου Καβαντά στο μέλλον και δίνω τον λόγο στον κύριο Καβαντά ως εισηγητή να ολοκληρώσει τώρα στο τέλος της συζήτησης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ε, να ευχαριστήσω και όλους τους προλαλήσαντες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή η έκθεση δεν πήγε στα σκουπίδια, ούτε μέσα σε ένα σιρτάρι. Ευχαριστώ λοιπόν όλους. Μου έκανε εντύπωση η προσπάθεια πολλών από εσάς ε, να παρασχέτε πραγματικά ε, καλές πληροφορίες. Να αναφέρω ένα δύο σημεία, όχι σημεία για τα οποία αναμένω απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα το 2012 ε, δεν, το 2013 συγγνώμη 100 θέσεις δεν μπόρεσαν να παρασχεθούν και 28 είναι γαλλόφωνες θέσεις. Το, λέω στη συμπατριώτησά μου να το πει στον Βασανπέιο που είναι ευρωβουλευτής ότι σε ένα κεντρικό γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα που περιλαμβάνει 1.200.000 διδάσκοντες, των οποίων 850.000 ε, ενεργοί διδάσκαλοι, μου κάνει εντύπωση που δεν μπορούμε να καλύψουμε τις θέσεις διδασκόντων ε, και για μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι προσπίζει τη γλώσσα της. Ο καθηγητής φιλοσοφίας του γιου μου, για παράδειγμα, ε, υπήρξε θύμα αυτής της δυσκολίας του συστήματος Επίσης 50 θέσεις ε, για Βρετανούς. Δεν νομίζω ότι θα πέθαινε η αυτοκρατορία. Αν καλύπτονταν αυτές οι θέσεις υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να πάει. Είναι αποτέλεσμα παρα... αμέλεια ουσιαστικά. 18 θέσεις λοιπόν είναι κενέ ε, για τους Γερμανούς για παράδειγμα επίσης. Για να ολοκληρώσω ήθελα να πω ένα πραγματάκι. Μου φαίνεται ότι από όλη αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια από όσο ξέρω από τους προκατόχους μου, αυτή η πρόταση της Κομισιόν, της οποίας ξέρω ότι καλή βούληση και του Επιτρόπου Σευκοβίτση πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να σκεφτούμε από νομική αψή το ενδεχόμενο να προσθέσουμε στη συνθήκη προσχώρησης ήδη από τώρα για τα επόμενα μέλη ως ένα πρόσθετο πρωτόκολλο κάτι που να λέει ότι υπάρχει υποχρέωση συμβολής των κρατών μελών ε, για τα παιδιά των όσων εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Λειτουργήμα. Δεν μπορεί το Βέλγιο να υφίσταται όλο το φόρτο, παρότι υπάρχει κάποιο οικονομικό όφελος. Δηλαδή να πάμε λίγο παραπέρα, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και πάλι ευχαριστούμε όλους τους προσκεκλημένους ε, πραγματογνώμονες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιστροφή στις χώρες σας. Συνεχίζουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη και περνάμε τώρα στην παρουσίαση της μελέτης ε, για την ε, εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καλωσορίζω τον κύριο Μπρουκ και την κυρία Ίνγε Φαντεν Έντε. Τι έχουμε εδώ. Η δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή προσπάθησε να διακριβώσει και να βρει με μία μελέτη, με μία αναζήτηση, έρευνα, διακόπτη η πρόεδρος. Ησυχία παρακαλώ. Καλό θα ήταν καθώς θα αποχωρείτε να μην συνομιλείτε και να διεξαγάγετε συζητήσεις εκτός εθούσης. Εντάξει. Θα θέλαμε να ακούσουμε τι συμβαίνει για τα διαφορετικά επίπεδα της εκμάθησης γλωσσών της γλωσσομάθειας και την συγκρισιμότητα σε σχέση με τα όσα γίνονται στις διαφορετικές διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο επιτυχές ήταν το εγχείρημα και τι έγινε. Έχει τον λόγο η κυρία Φαντενέντε ή ίσως ο κύριος Μπροκ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ε, thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ που μας προσφέρετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τις διακριβώσεις στα συμπεράσματα αυτής της μελέτης εξ ονόματος της ε, δικής σας ε, ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την εκπαίδευση και η μελέτη έγινε και από μένα και τους συναδέλφους και ένα ερευνητικό ίδρυμα με έδρα στην Ολλανδία. Μια σύντομη παρουσίαση, εισαγωγή της μελέτης πρώτα και μετά δύο λόγια για τα κυριότερα συμπεράσματα και τις συστάσεις που διατυπώνουμε. Και μετά την παρουσίαση θα υπάρχει και χρόνος για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ε, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ε, γλώσσες CEFR αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο για ε, την εκμάθηση γλωσσών στα κράτη-μέλη και να προαχθεί διαφάνεια και συνάφεια και συνεκτικότητα στην εκπαίδευση στις σύγχρονες ξένες γλώσσες στην Ευρώπη. Και δημοσιεύτηκε επίσημα το 2001. Το CEFR παρέχει ένα γενικό πλαίσιο που ε, λέει ποιες γλώσσες θα πρέπει να μπορούν να διδάσκονται ώστε να μπορούν να τις μαθαίνουν οι μαθητές στην πρακτική εφαρμογή και δημιουργώντας έτσι την κοινή βάση με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, εξετάσεις, μαθήματα που θα παρέχονται σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κράτη κτλ. Το CFR λοιπόν είναι μια με κατευθύνσεις προσέγγιση με έξι επίπεδα εκμάθησης γλωσσών από το α1 έως το C2 και κάθε επίπεδο εν δυνάμει μπορεί να περιγραφεί όσον αφορά τις επιδόσεις. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η συγκρισιμότητα μεταξύ των κρατών μελών μέσα σε μια κοινή προσπάθεια για την γλωσσική ε, εκπαίδευση αλλά και επίσης να έχουμε κοινέ προδιαγραφές σε αυτό το εγχείρημα. Οι συστάσεις του 2008 καλούν τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τις συστάσεις του CFR στα συστήματα στην εκπαίδευση και παιδεία των κρατών μελών να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την χρήση αυτού του κοινού πλαισίου και δεύτερον εξειδικευμένα μέτρα στο επίπεδο της πολιτικής ώστε να εκπαιδεύονται και να καταρτίζονται καθηγητές και δάσκαλοι και να προάγεται η αξιολόγηση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προήγαγε το CFR μέσα στο πλαίσιο της διαβίου εκπαίδευσης, μέσα στο πλαίσιο της παροχής και του διαβατηρίου ε, Europass που θα χορηγείται όσον αφορά τη, τη γλωσσική επάρκεια των ε, μαθητών. Ελήφθη υπόψη, ελήφθησαν υπόψη 14 ευρωπαϊκές χώρες και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα 45.000, επιδόσεων 45.000 μαθητών στην Ευρώπη υπό τους όρους του CFR. Με, αυτό το, με αυτά τα δεδομένα στόχος της μελέτης είναι να δοθεί η αξιολόγηση σε σχέση με τα σχολικά ε, εγχειρίδια και τις εξετάσεις. Να υπάρξει μια επισκόπηση τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την υλοποίηση του CFR, να παρασχεθούν συμπεράσματα, συστάσεις ε, και να ακολουθηθούν αυτά ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Για να δημιουργηθεί αυτό το ενιαίο πλαίσιο όσον αφορά την κοινή εφαρμογή μέλος, ε, όσον αφορά την μάθηση ξένων γλωσσών τίθεται το ερώτημα αν κατοχυρώνεται το CFR νομοθετικά σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, η χρήση στη δευτεροβάθμια, δευτεροβάθμια ε, εκπαίδευση με δυνατότητα να καλύπτονται οι ανάγκες στο συνολικό σύστημα ε, και τις ε, ανάγκες των μαθητών, σχολικά εγχειρίδια, κατάρτιση καθηγητών Τρίτον, οι χώρες ε, εξετάστηκαν σε σχέση με τις επιδόσεις τους ε, όσον αφορά την γλωσσική επάρκεια. Υπάρχει κάποια συγκλησιμότητα και συσχετισμός μεταξύ των όσων παρέχει το ECFR και τη αποδοτικότητα, των... της αποδοτικότητας των επιδόσεων. Προτού παρουσιάσω τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, δύο ε, λόγια για το τι έγινε. Επικεντρώσαμε την ανάλυση μας σε έξι κράτη-μέλη και έχουμε ένα είδο είδος ε, διπλώματος στο οποίο επικεντρωνόμαστε ανακριβώς κράτος μέλος ε, ε, που είναι η δυνατότητα πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση. Έχουμε λοιπόν τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά καθώς επίσης ε, και άλλες σύγχρονες γλώσσες όπως για παράδειγμα τα ισπανικά. Στην επιλογή των κρατών μελών λήφθη υπόψη αν χρησιμοποιεί το αυτό το πρότυπο και σε άλλες χώρες ή αν μπορεί να θεωρηθεί μια χώρα μόνο γλωσσική ή πολυγλωσσική λαμβάνοντας υπόψη τον, την ικανότητα να είναι να, έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται σε, σε μια άλλη γλώσσα επιπλέον οι κάτοικοι αυτής της χώρας. Επίσης και η γεωγραφική ισορροπία συμπεριλήφθηκε στην επιλογή των χωρών. Ε, είχαμε λοιπόν το στόχο να ε, ε, ερευνήσουμε σε βάθος εξειδικευμένα το τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες. Έγιναν συνεντεύξεις σε αυτές τις χώρες με εμπλεκόμενους. Είχαμε συνεντεύξεις και με τους παρόχους και συνεντεύξεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που διασφαλίστηκαν επίσης όσον αφορά τους εμπλεκόμενους. Εντάξει, αυτά είναι δεδομένα. Τώρα τα συμπεράσματα οι χώρες που χρησιμοποιούν το ECFR, CEFR σε διαφορετικό επίπεδο σήμερα ή πολλές φορές ε, δεν υπάρχει και καμιά αναφορά στο ε, CFR. Γενικά μπορούμε να αναφέρουμε όσο και περισσότερο χρησιμοποιείται στο νομοθετικό πλαίσιο ή στα μαθήματα το CFR, τόσο περισσότερο επηρεάζονται τα πράγματα όσον αφορά την εκπαίδευση των καθηγητών, τα σχολικά εγχειρίδια και τα συναφή. Έχουμε χώρες που έχουν ε, εμπεδώσει το CFR στην νομοθεσία τους. Κύριες προκλήσεις σε σχέση με την εφαρμογή τονίζονται δύο από αυτές ε, που θεωρούνται κυριότερες προκλήσεις. Ε, η απουσία εμπειρικών στοιχείων όσον αφορά την διασύνδεση του ε, ΚΕΠΑ και των επιδόσεων καθώς επίσης και τις εξετάσεις και άλλα έγγραφα σε σχέση με την πολιτική και δεύτερον την εφαρμογή του ΚΕΠΑ στις αίθουσες διδασκαλίες, διδασκαλίες που απαιτούν ειδικέ δεξιότητες σε κάποιες χώρες ε, η ε, Γαλλία, η Ολλανδία, η Σουηδία ε, έχουν, ανησυχούν για τη χρήση σε σχέση με το ΚΕΠΑ αν μπορούν να διασφαλιστούν οι αναγκαίες δεξιότητες για να ανταποκριθούν οι καθηγητές. Υπάρχει εδώ και απουσία δεδομένων. Δεν έχει γίνει κάποια μελέτη που να υπογραμμίζει τα επίπεδα διασύνδεσης μεταξύ ΚΕΠΑ και των εξετάσεων και των επιδόσεων στις εξετάσεις με βάση την προσέγγιση ΚΕΠΑ. Έγινε προσπάθεια να αναλυθεί η διασύνδεση σε σχέση με το πρόγραμμα εξετάσεων και το πρόγραμμα αξιολόγησης των επιδόσεων. Αλλά όπως έχει σημειωθεί δεν υπάρχει σαφής διασύνδεση που να κατοχυρώνεται νόμικα σε σχέση με τις εξετάσεις ε, και την προσέγγιση ΚΕΠΑ. Πρώτον επειδή δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός και διαφοροποίηση για τα διαφορετικά επίπεδα και οι περιγραφές των διαφορετικών επίπεδων είναι γενικόλογες, γενικού χαρακτήρα. Μία παρατήρηση. Κατά τα έτη κατά τα οποία εξελίχθηκε η προσέγγιση ΚΕΠΑ η στόχη του πλαισίου, η προσβασιμότητα, η περιγραφή των στόχων, το επίπεδο ε, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι επιδόσεις ε, στις ε, γλωσσικές δοκιμασίες. Κάθε επίπεδο σχεδόν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων και βλέπουμε ότι σε σχέση με εκείνους που διατύπωσαν γραπτός τις παρατηρήσεις τους ως επικρίσεις γενικότερα υπάρχει γενικότερη συμφωνία όσον αφορά την προσέγγιση του ΚΕΠΑ όσον αφορά την επίτευξη των μαθησιακών στόχων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βλέπουμε ότι τα επίπεδα είναι σχετικά συγκρίσιμα μεταξύ των έξι κρατών ε, που ε, λάβαμε ως σημεία αναφοράς και βλέπουμε ότι ε, στο δεύτερο επίπεδο έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Για την χρήση της προσέγγισης ΚΕΠΑ δείχνουν τα συμπεράσματα ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών που επελέγησαν υλοποιούν τηρούν αυτές τις υποδιαγραφές στις εξετάσεις στην Ουγγαρία, Αυστρία, Σουηδία και Ολλανδία. Οι εξετάσεις αυτές βασίζονται στην προσέγγιση και πά? Δεν συμβαίνει όμως αυτό στη Γαλλία, παρότι υπάρχει η διασύνδεση αυτή. Στην Σκοτία δεν υπάρχει μια τέτοια διασύνδεση. Ε, και τούτων λεχθέντων η διασύνδεση σε σχέση με τις, ε, ε, τη διδασκαλία σύγχρονων ξένων γλωσσών πρέπει να συμπληρώνεται με τα αναγκαία στοιχεία. Γενικά θα πρέπει να δούμε το πώς αναπτύσσονται τα θέματα αυτά στα σχολικά πλαίσια. Αν χρησιμοποιείται η προσέγγιση και στα μαθήματα και στα όσα διδάσκονται οι μαθητές σε σχέση και με τα εθνικά διδασκόμενα μαθήματα. Σε σχέση με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορούμε συναγάγουμε, του της Ευρώπης μπορούμε να συναγάγουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα χρήσης εγχειριδίων και σε κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κοινή κινήτρων που θα παρέχονται για να αναπτυχθεί αυτή η προσέγγιση. Εξετάζοντας την χρήση της προσέγγισης ΚΕΠΑ στην εκπαίδευση καθηγητών υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μαθήματα των οποίων την χάνουν οι καθηγητές προτού προσληφθούν. Χρησιμοποιούνται τα πλαίσια της προσέγγισης ΚΕΠΑ. Πρέπει να δούμε την εκπαίδευση καθηγητών ε, κατά τη διάρκεια της α, ε, ε, απασχόλησής τους στα σχολεία και την επιμόρφωση της οποίας μπορούν να τύχουν επειδή έχουν την ελευθερία να σχεδιάζουν τα μαθήματά τους οι καθηγητές σε πολλές χώρες, για παράδειγμα όσον αφορά την επιλογή του υλικού που θα διδάσκεται στους μαθητές όπως σχολικά εγχειρίδια, είναι δύσκολο να συναγάγει κανείς το συμπέρασμα αν χρησιμοποιείται όπως πρέπει αυτή η δυνατότητα από τους καθηγητές. Εξαρτάται από το, τη σπουδαιότητα που δίνεται στα κράτη ε, με, σε σχέση με τα μαθήματα που διδάσκονται και τη διδασκαλία τις οποίες την χάνουν ε, οι καθηγητές εξετάζουμε την δυνατότητα συσχετισμού του ε, ΚΕΠΑ και της ε, διδασκαλίας. Από τα διάφορα ε, δεδομένα όταν έχουμε τη γενική αξιολόγηση της, αξιολόγησης της προσέγγισης από τα κράτη-μέλη, η εξής αξιολόγηση μπορεί να προταθεί. Υπάρχει μια ομάδα πολύ υψηλών επιδόσεων στη Σουηδία και στην Ολλανδία. μια ομάδα υψηλών επιδόσεων στην Αυστρία, μέτριων επιδόσεων Ουγγαρία και Γαλλία και χαμηλών επιδόσεων ε, μεταξύ, ε, μεταξύ αυτών των χωρών το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σκοτία. Πρέπει επίσης να δούμε και τα επίπεδα ε, δεξιότητας που φαίνεται ότι βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα στις χώρες ε, με υψηλές επιδόσεις. Ο συσχετισμός όμως είναι ασαφής και πρέπει να, και άλλοι παράγοντες να ληφθούν υπόψη που διαδραματίζουν και αυτοί ένα ρόλο στις επιδόσεις. Αν η επίσημη γλώσσα για παράδειγμα χρησιμοποιείται ευρύτερα εκτός ε, ε, της ίδιας της χώρας ε, και τις ιδιομορφίες που συνεπάγεται αυτό. Επίσης και την, την αντίστροφη προσέγγιση. Χώρες με υψηλότερες επιδόσεις καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την δυνατότητα εφαρμογής των όσων προβλέπονται από την προσέγγιση ΚΕΠΑ. Γενικά θα πρέπει να δούμε και τους ε, παρόχους ε, ε, κατά πόσον οι επιδόσεις διασφαλίζονται και μέσω των πιστοποιητικών και σε σχέση και με το επίπεδο το οποίο επιτυγχάνεται και κατά πόσον συνειδητοποιούν οι καθηγητές τις ανάγκες που υπάρχουν μέσω της εκπαίδευσής τους. Παρότι είναι χρήσιμα τα εγχειρίδια και αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, παρόλα αυτά ο περίπλοκος χαρακτήρας που έχει η προσέγγιση ΚΕΠΑ επιβαρύνει πολλές φορές τα πράγματα. Υπάρχουν, ε, ε, ε, υπάρχει διεκδίκηση, υπάρχει το αίτημα να απλουστευτεί αυτό το πλαίσιο για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα πρέπει εδώ να διασφαλίζεται η διαφάνεια ώστε να εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες των ευκαιριών που θα παρέχονται ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να, έχουμε, να υπάρχει πρόσβαση στα πανεπιστήμια και να αυξάνεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ε, οι όσοι ε, αποφυτούν από αυτά τα μαθήματα. Η προσέγγιση ΚΕΠΑ ε, θέλει να διευκολύνει τη συγκρισιμότητα αυτών των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών και να καθίσταται περισσότερο συγκρίσιμη η προσπάθεια από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε τις ε, εξής συστάσεις που υποβάλλουμε. Η σύσταση υπαριθμών 1 θα πρέπει η ΚΕΠΑ από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρυνθεί ω εργαλείο για την ε, προώθηση αυτή τη προσπάθεια. Υπάρχει η προσέγγιση ΚΕΠΑ εδώ και πάνω από 10 χρόνια και πολλέ εξέλιξει έχουν σημειωθεί. Όμω ε, στην εφαρμογή θα μπορεί να υπάρξει μια νέα προώθηση και γι' αυτό συνιστούμε να αναπτύξουμε περισσότερο την ε, δυνατότητα αυτή που ανέφερα πιο πριν, συμπεριλαμβάνοντας και περισσότερες χώρες και περισσότερες γλώσσες σε αυτή την προσπάθεια. Όχι μόνο τις δύο, ε, τις περισσότερο ε, διαδεδομένες γλώσσες όσον αφορά την εκμάθηση, αλλά και το επίπεδο της εκμάθησης δεύτερης γλώσσας θα πρέπει να συμμεριζόμαστε ε, την πείρα και την εμπειρία στα κράτη-μέλη ώστε να είμαστε περισσότερο δραστήριοι στις ε, δράσεις που θα αναλαμβάνουμε και ε, επισημένοντας το επίπεδο ικανότητας μεταξύ των όσων εμπλέκονται. Θα πρέπει εδώ να έχουμε μια ενιαία δυνατότητα υποβολής των όσων σημειώνονται στα κράτη-μέλη τρίτων και περισσότερο θα πρέπει ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus ε, ΣΥΝ να παρέχουν δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα και δυνατότητες προαγωγής του ευρωδιαβατηρίου Europass και ένας συντονισμός ευρωπαϊκός με μια παρόμοια βάση θα πρέπει να οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα με αυτή τη δυνατότητα. Δεύτερη σύσταση να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ των συστημάτων ΚΕΠΑ και των χωρών. Διασύνδεση μεταξύ συστημάτων και του ΚΕΠΑ από τις χώρες. Παρότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα μαθησιακά αποτελέσματα των ε, ξένων γλωσσών που διδάσκονται, η σύνδεση αυτή δεν αναγνωρίζεται από τα άλλα κράτη η σύνδεση αυτή δεν αναγνωρίζεται από άλλα κράτη-μέλη, εν λόγω αναγνώριση δεν είναι καθεαυτή απαραίτητη. Όταν όμω τίθεται το ζήτημα αμοιβαία εμπιστοσύνη στα προσόντα και τα πιστοποιημένα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διαδικασίε που εφαρμόζονται θα πρέπει να είναι τέτοιε ώστε να συνδέονται τα συστήματα αυτά στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών όσον αφορά την ΚΕΠΑ. Δεν είναι μόνο τεχνικού χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί δυνατότητα να προαχθεί η πολιτική κοινωνική συζήτηση αρχές θα μπορούσαν για παράδειγμα να είναι οι εξή. Συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής εμπειρογνωμόνων, διδασκόντων στα σχολεία, εκδοτών, αξιοποίηση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, θέσπιση ενός κοινού σχεδίου ε, που θα μπορούσε να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερη σύσταση να διευκολύνουμε την εμπλοκή άλλων χωρών στη διασύνδεση σε σχέση με την ε, ε, μάθηση ξένων γλωσσών. Κύριο ερώτημα είναι ε, αν ε, μπορούν να υπάρξουν τέτοιες δυνατότητες ε, και να τρίτον να δώσουμε τη δυνατότητα αύξησης της πραγματικής χρήσης του ΚΕΠΑ ώστε να υπάρχει διασύνδεση σαφής μεταξύ των εθνικών συστημάτων και του ΚΕΠΑ ώστε να υπάρξει ένα σύστημα μεταρρύθμισης δράσεων μεταρρυθμιστικών. Τρίτη σύσταση, να αυξηθεί η πραγματική χρήση του ΚΕΠΑ στα σχολεία γιατί όπως είδαμε η χρήση του ΚΕΠΑ σε βασικό επίπεδο <clears throat> ενισχύεται από πολιτικές δράσεις υψηλού επίπεδου, όπως η ενσωμάτωση του ΚΕΠΑ στην ομοθεσία ή η χρήση στον καθορισμό των εθνικών προγραμμάτων σπουδών. Και επιπλέον ε, απαιτούνται περαιτέρω δράσεις ώστε να παρακινηθούν οι διδάσκοντες και οι εκδότες να χρησιμοποιούν το ΚΕΠΑ ευρύτερα. Γι' αυτό συνιστάται η δημιουργία αξιοπιστία και καλύτερη εφαρμογή του πλαισίου σε εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας, κάνοντα χρήση τη εμπειρία και των συζητήσεων με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χρησιμοποιώντας τι συμβουλές εμπειρογνωμόνων και το εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιπρόσθετα για τους σκοπούς τη σαφέστερης χρήση το ΚΕΠΑ πρέπει να ε, κατοχυρώνεται, να εντάσσεται στα εθνικά προγράμματα σπουδών και έτσι στα ειδικά προγράμματα σπουδών ξένων γλωσσών, ώστε να ιδρωθεί πλήρω η εκμάθηση αυτών και η προσέγγιση που προσανατολίζεται στην ανάληψη δράση. Ε, επιπλέον, ε, χρειάζεται έρευνα και εποπτεία. Θα ήταν αναγκαίο να υπάρχει υποστήριξη και κατευθυντήριε γραμμέ, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε δυνατότητε πιο αυξημένου επίπεδου μάθησης να, υπάρξει επίσης, να υπάρξουν κίνητρα ε, για να ε, μπορέσουν ε, να γνωρίζουν τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι διδάσκοντες μπορεί αυτό να γίνει δίνοντας κίνητρα για παράδειγμα ανταλλαγής μεταξύ, ανταλλαγών μεταξύ αυτών των δυνατοτήτων και να διευρυνθεί η δυνατότητα με μια πιο δραστήρια, με ένα πιο δραστήριο προσανατολισμό. Τελευταία σύστασή μας Παρότι η μελέτη καλύπτει ένα ευρύτερο πλαίσιο, πολλά θέματα γύρω από το ΚΕΠΑ παραμένουν ασαφή. Αυτά αφορούν κυρίως κοινωνικά πολιτικά ζητήματα που συσχετίζονται με την εκμάθηση γλωσσών και γι' αυτό συνιστούμε την περαιτέρω μελέτη των εξή θεμάτων. Ποιες είναι οι αναδυόμενες, ανερχόμενες γλώσσες και πώς μπορεί το ΚΕΠΑ να είναι αρκετά ευρύ ώστε να καλύψει μη ευρωπαϊκές γλώσσες όπως τα κινέζικα ποιες είναι οι επιπτώσεις ενός ευρωπαϊκού δίκτυ γλωσσών στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη γλώσσα. Καθιέρωση ενός δίκτυ που αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για περαιτέρω ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου, όμως δεν πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο περιορισμένη εστίαση στην εκμάθηση γλωσσών. Και ένα τρίτο θέμα. Πώς μπορεί το ΚΕΠΑ να χρησιμοποιηθεί, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενδυναμωθεί ε, η θέση των λιγότερο διαδεδομένων μειονοτικών γλωσσών και να υπάρξει ένα υπερεθνικός ε, φορέας ή όργανο που θα δημιουργηθεί ή μια συμβουλευτική ομάδα στις χώρες εκείνες ε, που να επανεξετάζουν την αντιστοίχηση που θα έχει επιτύχει κάθε μια μεταξύ των πολιτικών εκμάθησης γλωσσών και του ΚΕΠΑ. Αυτό το υπερεθνικό όργανο μπορεί να λειτουργεί ω πλατφόρμα για ανταλλαγή εμπειριών για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, παροχή πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών, δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης ε, στην αντιστοίχηση μεταξύ προσόντων ε, στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Και συνοψίζουμε, το ΚΕΠΑ θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για να αυξηθεί η ε, ικανότητα στις ξένες γλώσσες και να αυξηθεί έτσι μια δραστήρια προσέγγιση στην εκμάθηση γλωσσών. Χρησιμοποιείται το ΚΕΠΑ στα κράτη-μέλη σε διαφορετικό βαθμό εκάστοτε όσον αφορά την κατοχήρωσή του σε νομικά έγγραφα και νομικά πλαίσια, στη χρήση σε σχολικά εγχειρίδια, καθώς επίσης και στην κατάρτιση και εκπαίδευση ε, του ε, καθηγητικού προσωπικού. Πρέπει να υπάρξει μια ενδυναμωμένη προσπάθεια ενδυναμώνοντας ε, τη διασύνδεση των διαφορετικών επιπέδων και περαιτέρω αναπτύσσοντας το ΚΕΠΑ και απλουστεύοντάς το. Σας ευχαριστώ. Vielen herzlichen σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και είμαι, και σίγουρη, ότι θα ασχοληθούμε και στο μέλλον. Θα ασχοληθούμε και στο μέλλον με αυτό. Τώρα, όποιο θέλει να ε, λάβει τον λόγο, αν εσεί θέλετε να παρέμβετε, έχετε τον λόγο. Δύο λόγια μόνο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Επιτρέψτε μου να τονίσω και να πω ότι είμαι υπερήφανος ότι κατά τη διάρκεια της Σλοβενικής Προεδρίας η πρόθεση αυτή που δόθηκε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πολυγλωσία, στο πολυγλωσσικό καθεστώς ήταν κάτι θετικό και με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι μπορούμε να δρέψουμε τους πρώτους καρπούς ως πρώτα αποτελέσματα σήμερα. Να τονίσω σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη το ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και αυτά τα νεότερα κράτη-μέλη σε αυτή τη μελέτη, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τα διάφορα θέματα και σε σχέση με αυτά τα κράτη. Και υποστηρίζω τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που μας παρουσιάσατε. Και επίσης μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ακριβώς από το πώς θα προαγάγουμε την αμοιβαία κατανόηση και πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε και τις γλώσσες. Η γνώση γλωσσών μπορεί να ε, οδηγήσει στην προαγωγή της αμοιβαία κατανόησης. Είναι ένα αναγκαίο στοιχείο. Έχει τεράστια σημασία λοιπόν να ξέρει κανείς να μαθαίνει άλλες ξένες γλώσσες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα των γειτόνων του. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει που θέλει να πάρει το λόγο. Όχι λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βαν Κρόκ και Βαν Έντε και νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα, αυτό το κείμενο ε, πραγματικά θα μας δώσει πολλά ραθίσματα και, πολλά, και ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκλογική μας περιφέρεια ώστε οι πολίτες να καταλάβουν τη σημασία της εκμάθησης των ξένων γλωσσών και να μπορέσουν να ρίξουν μια ματιά και οι καθηγητές. Εγώ θα έχω μια συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας γιατί η χώρα μου αποφάσισε να είναι δίγλωση. Να έχουμε δηλαδή και τα γαλλικά, γερμανικά και γαλλικά, όχι βεβαίως ε, ε, από αύριο, αλλά μελλοντικά. Γιατί όχι λοιπόν, θα μπορούσαμε να το προσπαθήσουμε. Πολλοί στη Γερμανία πιστεύουν ότι οι άνθρωποι μας στο μιλάνε γαλλικά, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Τώρα όμως θα προσπαθήσουμε πραγματικά να το κάνουμε, να το πραγματοποιήσουμε. Άρα λοιπόν το εργαλείο αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο στην κυβέρνηση και τώρα θα ήθελα να πω ότι λύεται η συνεδρίαση. Τώρα έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών. Όσοι, όλοι όσοι δεν ε, ε, ανήκουν στους συντονιστές παρακαλώ να αποχωρήσουν.